έχει ε, θεσμοθετήσει 7 blending facilities. χρησιμοποιώντας και την εξωτερική συνεργασία. Ε, ε, στα facilities αυτά υπάρχουν, υπάρχει ένα μείγμα επιδοτήσεων ε, με μη δανειακούς ε, πόρους που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μετά, σε επίπεδο ε, έργου, project, κάθε μορφής πόρη αναμειγνύονται. Γίνεται αυτό το blending δηλαδή και προωθούνται προς συγκεκριμένα προγράμματα. Για να απεικονίσουμε καλύτερα το θέμα αυτό, έχω προετοιμάσει αυτό το μικρό γράφημα όπου βλέπετε σε μια ε, διαδικασία blending αρχικά ε, θα ε, πρέπει να υπάρξει το αίτημα από την ετούμενη χώρα και μετά έχουμε τους κοινοτικούς ενωσιακούς πόρους που μπορούν να ακολουθηθούν από ιδιωτικούς πόρους, αλλά κυρίως και από πόρους δημοσίων ε, οργανισμών. Μπορεί να είναι η KFW, μπορεί να είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, και Ανάπτυξης κτλ. Εκεί μπορεί κανείς να προσθέσει και ε, ας πούμε όπως άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα Ανάπτυξης κτλ. Επιπλέον, μπορεί κανείς να ε, έχει και ιδιωτικούς ε, και ιδιώτες ε, επενδυτές ή εμπορικούς επενδυτές που μπορούν να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα προγράμματα σε συνεργασία με τις τοπικές περιφερειακές κυβερνήσεις. Νομίζω ότι πρέπει κανείς να καταλάβει ότι από το 2007, να συνειδητοποιήσει, από το 2007 οι, αυτές οι 7 facilities έχουν ε, λειτουργήσει. Είναι η LIFE, είναι η ITF, είναι η Neighborhood Investment ε, Facility για την ε, Κεντρική Ασία και για την Ασία γενικότερα και μέσω αυτών έχουν μπει σε πάγια 1,2 δισεκατομμύρια ε, βάσει των οποίων έχουν ε, προκύψει επιπλέον χρηματοδότηση της τάξης των 32 δισεκατομμυρίων. Ε, είναι σε δάνεια, επιδοτήσεις και equities είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβει ε, αυτό η υπόψη του κανείς, κυρίως δε, ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική, το αρχικό πρόσωπο ήταν μάλλον μικρό, αν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι μικρό το ένα δις. Λοιπόν, εδώ σας δείχνω ένα άλλο χάρτη, ένα άλλο γράφημα, ε, για να δείτε ότι συνολικά από το 2007 έχουμε χρηματοδοτήσει 168, 170 projects ξεκινήσαμε το 2007 με μία απλή ιδέα. Το 2008 δημιουργήσαμε την Neighborhood Facility, μετά ε, από ένα χρόνο την Life και την IFCA και το 2012 ε, ξεκινήσαμε ήδη την, ε, το επενδυτικό εργαλείο για την Καραϊδική κλπ. Βλέπετε εδώ το σύνολο της χρηματοδότησης και τον καταμερισμό σε, ενωσιακό και μη, σε ενωσιακή και μη ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα ήθελα να σας δείξω, να σας πω ότι το blending ε, χρηματοδοτεί συγκεκριμένα προγράμματα και ε, θέλει να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα τα αποτελέσματα είναι σαφή και προφανή. Εγώ έχω δώσει κάποια παραδείγματα εδώ, ας πούμε στην Ικαράγουα. Θα χρηματοδοτήσουμε ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου η αύξηση σε πόσιμο νερό από το 72% του πληθυσμού θα φτάσει στο 75% σε 15 πόλεις. Στο Μαρόκο Έχουμε στην, ε, την χρηματοδότηση του μεγαλύτε, της μεγαλύτερης ηλιακής εγκατάστασης ε, στην Βόρεια Αφρική που θα μειώσει την εξάρτηση από την ε, εισαγωγή ενέργειας και θα, θα, θα, περικόψει 250.000 τόνους διοξιδίου του άνθρακος. Στη Δυτική Αφρική 1.300 χιλιόμετρα γραμμές μετάδοσης που θα, συν, που θα βοηθήσουν 60.000 νοικοκυριά να ενωθούν με το ηλεκτρικό ρεύμα. Στην ε, Ανατολική Αφρική επίσης, ε, στην, ε, στο, στην, στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας επίσης. Τώρα, ποιους τομείς καλύπτουμε. Καλύπτουμε κυρίως τους τομείς ενέργειας και ακόμα περισσότερο τον τομέα της μεταφοράς. όλο και περισσότερη χρηματοδότηση πηγαίνει προς το νερό και την αποχέτευση ένα αρκετά μικρό ποσοστό ακόμα αφορά στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που παρόλα αυτά φτάνει το 11%. 5% αφορά κοινωνικές δαπάνες, μπορώ να σας πω γιατί ο μηχανισμός ανάμιξης, ο blending mechanism δεν είναι ο πλέον προσήκον για τη χρηματοδότηση κοινωνικών έργων ε, και έχουμε για την πληροφορική και την ε, ε, επένδυση στην πληροφορική 3%. Όσον αφορά τώρα τα είδη επενδύσεων, ε, χρηματοδοτούμε κατά 41% άμεσες ε, επενδύσεις. Το 1 τρίτο περίπου, 30% αφορά την τεχνική ε, βοήθεια, την διαχείριση, τις ε, μελέτες για περιβαλλοντική επίπτωση, κοινωνική επίπτωση των έργων κτλ. Ε, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 19% αφορά την την, ε, τις, ε, τα επιτόκια, κυρίως αν μιλάμε για την ε, ΑΕΦ και 4% πηγαίνει στο κεφάλαιο κινδύνου και 3% στις εγγύησεις. Εάν θέλουμε να δουλέψουμε χέρι-χέρι με τον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει οπωσδήποτε στα δύο αυτά κεφάλαια να προχωρήσουμε εντονότερα από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα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 ε, έλεγα προηγουμένως ε, ότι η ατζέντα που έχουμε για την συνεργασία ε, θέλει, ζητάει συνεργασία με όσο γίνεται περισσότερους φορείς έτσι ώστε και η επίπτωση και η αποτελεσματικότητα της ενωσιακής βοήθειας να είναι μεγαλύτερη. Θέλουμε μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα και μεγαλύτερη συνοχή. Και εγώ θα προσπαθήσω να σας πω ότι ε, έχουμε επιτύχει βελτίωση της ε, βοήθειας που δίνουμε. Επίσης, ε, μέσω του blending μειώνεται το κόστος της συναλλαγής, το διοικητικό κόστος για τις συμμετέχουσες χώρες και επίσης απελευθερώνει κεφάλαια και πόρους για άλλα επιπλέον προγράμματα. Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας blending είναι ότι εμείς έχουμε συνενώσει τέσσερις διαφορετικούς κόσμους, ε, Ευρωπαίους και μη Ευρωπαίους πρωταγωνιστές για την βοήθεια, τράπεζες κτλ. από τις περισσότερες πλευρές του κόσμου και επίσης δύο κόσμους που ήταν χωριστοί μέχρι τώρα. Τον κόσμο των δονητών, των δωρητών και τον κόσμο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με, έχοντας βεβαίως ε, τον ίδιο στόχο, δηλαδή την ανάπτυξη των ενωσιακών ε, στόχων. Επομένως, θα μπορούσα να είπω ότι η αύξηση της αποτελεσματικότητας είναι το κύριο, το μεγάλο κλειδί και η ανάμειξη, η blending έχει καταλήξει σε μεγαλύτερη συνεννόηση και συνέργεια μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και δωρητών καθώς και την καλύτερη ταύτιση και προετοιμασία των σχεδίων και γι' αυτό υπήρξε η καλύτερη συνεργασία. Τώρα για να συνοψίσω. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ανάμιξη, το blending δεν αφορά μόνο τη μόχλευση. Υπάρχει, υπάρχει και αυτή και το τόνισα σε προηγούμενη διαφάνεια όπως σας είχα αποδείξει ελπίζω ότι πρόσθετες, πρόσθετη δημόσια και ιδιωτική πόροι καταλήγουν σε μεγαλύτερο αποτέλεσμα αλλά υπάρχει και μη χρηματοπιστωτικό θέμα με το blending βελτιώνουμε τη βιωσιμότητα και την ταχύτητα εφαρμογής των σχεδίων και υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία από τις συμμετέχουσες χώρες. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει και μία πτυχή πίστοσης σε όλα αυτά. Τέλος τέλος δε, είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε ότι όσα κάναμε και όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε ευθυγραμμίζονται με, τη, με τα ενωσιακά προγράμματα και τους ανεπτυξιακούς στόχους που έχουν τεθεί και περιφερειακά και γενικά. Θα ήθελα τώρα να σας διαβεβαιώσω για την επιλογή των σχεδίων ή προγραμμάτων πρέπει να αναφέρουμε ορισμένα σημαντικά πράγματα, να μην γίνει στρέβλωση της αγοράς και με τις δωρεές να υπάρξει προσθετικότητα. Κάναμε μία ανάλυση γεωγραφική και θεματική με τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις περίπτωση την περίπτωση για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε λάβει πράγματι υπόψη μας τα επίσημα περιφερειακά κριτήρια και τη συνέπεια τη συνοχή καθώς και όλα τα τεχνικά προβλήματα όπως το όφελος που έχουν όλα αυτά, τη μόχλευση και τη βιωσιμότητα. Να σας εξηγήσω. Προς το παρόν, και νομίζω οι αριθμοί το δείχνουν, κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να στηρίξουμε δημόσια σχέδια επενδύσεων 90% αλλά επίσης είπα ότι το blending μας δίνει και τη δυνατότητα να κινητοποιήσουμε και τις ιδιωτικές επενδύσεις μέσω καινοτόμων δημοσιονομικών ή χρηματοπιστικών εργαλείων όπως τα παρακινημένα κεφάλαια και οι εγγυήσεις των επενδύσεων. Χρειάζονται να γίνουν κι άλλα βέβαια άλλα. Θέλουμε όμως να βελτιωθεί, να αυξηθεί το bullending για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε δημιουργήσει μια ολόκληρη ενωσιακή πλατφόρμα σε συνεργασία με κράτη, υπηρεσίες της Κομισιόν, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιωθεί ό,τι κάναμε μέχρι τώρα και η μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση για το, για το πρόγραμμα ενίσχυσης της πολιτικής γειτονίας απέδειξε ότι υπάρχει καλύτερη συνεργασία έτσι. Αναθεωρούμε αυτή τη στιγμή συστηματικά όλα, όλες τις διευκολύνσεις και τα εργαλεία με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε και επειδή αφού είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλω να τονίσω ότι αυτό συμμετέχει και τεχνικά και στο σχεδιασμό της στρατηγικής ή πολιτικής. Και για τέταρτη φορά τέλος έχουμε δύο τεχνικές ομάδες. Την ένα όπου συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα και τις διαδικασίες των διαφόρων μηχανισμών bullending τονίζουμε ιδιαίτερα τα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε και τις βέλτιστες πρακτικές και αναθεωρούμε τη δομή της διακυβέρνησης και την ομάδα 2, τεχνική ομάδα 2, για να υπάρξει ένα πλαίσιο που να βασίζεται στα αποτελέσματα και να μετράει την αποτελεσματικότητα και την προσθετικότητα των δωρεών τουλάχιστον και αυτό μάλιστα με τρόπο τυποποιημένο ώστε να υπάρξει ένας συνεπής μηχανισμός που να μας επιτρέπει, ανάλυσης που να μας επιτρέπει να απαντήσουμε στα προβλήματα που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των δύο τεχνικών ομάδων αναμένονται τον Ιούνιο και θα συζητηθούν στην ομάδα πολιτικής. Σας κατευχαριστώ για την ε, υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Σοφή Σιρτέν από την Παγκόσμια Τράπεζα. Έχει εργαστεί σε διάφορες περιφέρειες και ε, παραρτήματα ε, της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η κυρία Σιρτέν θα μας δώσει την άποψη Παγκόσμιας Τράπεζας για την αποτελεσματικότητα της ναι. βοήθειας και την αναπτυξιακή συνεργασία. Έχετε το λόγο. Thank you. Let me just take a minute to find my presentation. I suppose it's somewhere here. Μια στιγμή να βρω την τοποθέτησή μου στο μηχάνημα. So as it's being loaded, um, let me explain the... Φορτώνει. Να σας πω τι στόχο έχω να σας δώσω μια γενικότερη θεώρηση και κάποιες σκέψεις για το πώς μπορεί να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας. Θα σας δώσω λίγο το πλαίσιο. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό το όλο θέμα. Και μετά θα σας πω τι φρονεί η Παγκόσμια Τράπεζα και πώς θεωρούμε εμείς ότι μπορεί να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας και θα κλείσω με ε, μερικές προτάσεις και μερικές σκέψεις για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το πλαίσιο γενικότερα, ακούσατε από τον προλαλήσαντα, αλλά και τις Προεδρούς, ότι το 2015 ήγγηκε η ώρα που είχαμε θέσει ως στόχο για ...την αναπτυξιακή βοήθεια του στόχου της χιλιετίας. Η διεθνή κοινότητα αναπτυξιακή βοήθεια τώρα προβληματίζεται για ένα νέο πλαίσιο και πώ θα χρηματοδώσει τι ε, ε εναπομείνασε τεράστιε όμω ανάγκε και τις βασικέ προτεραιότητε. Βλέποντα εδώ τη γραφική παράσταση, βλέπετε ότι η κρατική αναπτυξιακή βοήθεια είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα όλων των χρημάτων. Λιγότερο από το 1% ε, όλων των ε, χρηματικών ροών που πηγαίνουν ε, προς την αναπτυξιακή βοήθεια και η μερίδα του λέοντος είναι από τον ιδιωτικό τομέα με διάφορους τρόπους. Αυτό τονίζεται περισσότερο από το γεγονός ότι πέρσι λόγω της κρίσης έχουν μειωθεί οι πόροι από τη δημόσια βοήθεια γιατί μειώνουν τη χρηματοδότηση με περικοπές οι διάφορες χώρες. Ακόμα και προσπαθούν να δίνουν αρκετά χρήματα, παραμένουν, ε, υπολείπονται κατά πολύ των στόχων που είχαν ε, ε, αποφασίσει στο Μόντερεϊ. αν θυμάστε. Θα πρέπει λοιπόν από το νέο πλαίσιο, μετά το 2015, να αλλάξει η κατάσταση. Αν κοιτάξετε τις μεγαλύτερες ζωές λοιπόν από τον ιδιωτικό τομέα, τι διαπιστώσετε. Είναι πάρα πολλοί μεταβλητές από χώρε με μέσο εισόδημα έπεσαν ε, μέχρι και κατά 30% ε, στο ζενήθ της κρίσης. Επίσης, στις λιγότερο ρεπτυγμένες οικονομίες πηγαίνουν πολύ λιγότερα χρήματα πλέον και οπωσδήποτε ανεπαρκεί για να καλύψουν ε, τις ανάγκες τους. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού να ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθηθούν αυτές οι χώρες από το 2015 και μετά για να μεγιστοποιηθεί ε, όσο γίνεται η ε, ωφέλεια από τη δημόσια βοήθεια. Αυτό θα ήθελα να σας εξηγήσω λοιπόν πώς πιστεύουμε ότι θα πιάνουν καλύτερα τόπο ε, τα ευρώ ή τα cents όλα. Λοιπόν, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, η δημόσια, ε, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, να πιάνει το όπως είπαμε και επίσης θα πρέπει να υπάρξει μία μόχλευση, μία ανάμνηξη ε, ε, με άλλους πόρους ιδιωτικούς. Η υπόλοιπη παρουσίασή μου λοιπόν αφιερωμένη στο πώς θα φτάσουμε εκεί. Πώς θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της βοήθειας η διεθνής κοινότητα έχει επαρελειμμένα συναντηθεί για αυτό το θέμα. Μοντερέι, Παρίσι, Άκρα και το 2011 ήταν η τελευταία φορά. Είναι πολύ λογικά αυτά που ζητούμε σε ένα πλαίσιο ε, θα πρέπει να ενταχθούν για να παρακολουθούμε την πρόοδο. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο και τι αναγνωρίζει. Είναι πιο αποτελεσματική η βοήθεια όταν γίνεται κτήμα των κρατών. Δηλαδή, ε, όταν ευθυγραμμίζεται με τις εθνικές κρατικές στρατηγικές για να μπορούν να ε, το αγκαλιάσουν αυτό οι κυβερνήσεις και να το εφαρμόσουν. Το περίφημο ownership. ownership να μειωθεί το γραφειοκρατικό κόστος και η διαδικασία, η συνεργασία με τους διάφορους εταίρους, ε, να βασιζόμαστε στα διάφορα συστήματα των ε, ε, κρατών και να υπάρχει μια διμερή συνεργασία των δωρητών. Επίσης, είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα και βάσει αυτό να κρίνουμε και να είμαστε και υπόλογοι των αποτελεσμάτων. Όπως βλέπετε από αυτή τη γραφική παράσταση παραμένουν πάρα πολλοί έγκυρες αυτές οι προτάσεις και στην ημερήσια διάταξη για όλους που ασχολούμαστε με την αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά δεν αρκούν αυτά όλα. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. Να πιάνουν τόπο τα χρήματα. Πώς μετράμε λοιπόν αυτό το στόχο. Θα πρέπει να, ακριβώς να εστιάζουμε στα αποτελέσματα. Από το αποτέλεσμα κρίνουμε κάθε φορά, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η δυνατότητα να καθορίσει κανείς τους επιθυμητούς στόχους. Πού θέλουμε να φτάσουμε, τι θέλουμε να επιτύχουμε μαζί με τις χώρες πελάτες μας για να έχουμε σαφείς στόχους που μπορούμε και να ελέγχουμε, να είναι μετρήσιμοι και να είμαστε και υπόλογοι. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο έργων, προγραμμάτων, θεσμών, στρατηγικών, χωρών ή ακόμα και στόχων που έχουμε θέσει ως διεθνής αναπτυξιακή κοινότητα. Επίσης πιστεύουμε ότι χρειάζεται να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται περισσότερο το feedback, αυτά που μας αναφέρουν οι ενδιαφερόμενοι για να αξιολογούμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Ε, τα μέσα, οι μεθοδολογίες, οι πολιτικές που προσφέρονται σε ένα δεδομένο περιβάλλον για να φτάσουμε στους επιθυμητούς στόχους. Όλα αυτά είναι κρίσιμα. για να μπορέσουμε όσο γίνεται να συμβουλεύουμε καλύτερα τις χώρες. έχουμε αναπτύξει στην Παγκόσμια Τράπεζα αυτό που ονομάζουμε η επιστήμη της παροχής, science of delivery. Ε, δηλαδή πώς εφαρμόζεται κάθε βοήθεια, να υπάρχει μια τεχνογνωσία, ένα savoir-faire εφαρμογής και υλοποίησης. Δηλαδή να βοηθούμε να συνοδεύουμε τις χώρες όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το καθένα από αυτά για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας γιατί κάθε φορά έτσι αυξάνεται η λογοδοσία όχι μόνο των δωρητών αυτών καθ' αλλά και των κυβερνήσεων προς τους πολίτες τους. Ε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Υπάρχουν και ε, ειδικέ επιμέρους ενότητες και κλάδοι που μπορεί κανείς να μετρήσει το ευεργέτημα και το όφελος της περισσότερης διαφάνειας, ακόμα και σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εδώ. Να δημοσιεύουμε περισσότερο τα όσα κάνουμε εμείς ως δωρητές, να ενθαρρύνουμε και τους αποδέκτες να τα διαβιβάζουν αυτά, να ενημερώνουν τους πολίτες και να ενισχύουμε το ρόλο των τελικών δικαιούχων στις χώρες. Να συμμετέχουν από την αρχή στο σχεδιασμό των όσων κάνουμε εμείς, αλλά και να μας αναφέρουν ε, τις εμπειρίες τους για να έχουμε ένα feedback κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της υλοποίησης των προγραμμάτων και χρειαστεί τα προγράμματα αυτά να διορθώνονται στην πορεία. Ένα άλλο μέσο που χρησιμοποιούμε μαζί με άλλους ε, δωρητές είναι ε, η γεωχαρτογράφηση. Geomapping. Εδώ βλέπετε το παράδειγμα του Μαλάουι. Είναι χρήσιμο για τους δωρητές να γνωρίζουν ε, που υπάρχουν ελλείψεις, που υπάρχουν επικαλύψεις. Εδώ θα έχετε στοιχεία αν μπείτε στο site ε, ενημερώνεται το site αυτό σε πραγματικό χρόνο από τις ομάδες που συμμετέχουν στα έργα αυτά. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη προϋπόθεση σε αυτά που λέω. Αν οι κυβερνήσεις ε, συνειδητοποιήσουν ότι όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς, χωρίς καλές στατιστικές. Μπορεί να έχετε ό,τι προβλήματα θέλετε, ό,τι προγράμματα θέλετε, χρηματοδότηση. Αν δεν έχετε σωστές στρατηγικές δεν μπορείτε στατιστικές συγγνώμη, να ε, εκτιμήσετε ένα πρόγραμμα. Σε πολλές χώρες υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, ιδιαίτερα σε φτωχές χώρες με τις στατιστικές. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Στην Νότια Ασία και την Υποσαχάρη Αφρική, κάτω από το 2% του πληθυσμού ζει σε χώρες που έχουν ενημερωμένες ε, στατιστικές για γεννήσεις και θανάτους. Πάνω από τις μισές χώρες στην Υποσαχάρη Αφρική δεν έχουν κάνει έρευνα την τελευταία πενταετία στα νοικοκυριά. Και είναι κρίσιμες αυτές οι έρευνες για να συλλέξεις πληροφορίες, για να δεις ποια είναι τα προβλήματα και οι ανάγκες του πληθυσμού. Πριν από ένα μήνα λοιπόν υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεννόησης με ε, διάφορες ε, αναπτυσσόμενες χώρες ε, και σκοπός μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα. Έχουμε τώρα στην μόχλευση. Okay. Συνδυασμός λοιπόν διαφόρων πηγών. Εγχώριες πηγές, δεν είναι πάντα ο ιδιωτικός τομέας. Υπάρχουν και εγχώριες ε, που μπορούν να μοχλευθούν καλύτερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, ε, καταφέρνουν έτσι οι χώρες να εξαρτώνται λιγότερο από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά και να ε, ε, έχουν ε, μεγαλύτερο έλεγχο και να είναι κτήμα τους αυτή η διαδικασία. Βλέπετε εδώ σε αυτό τον πίνακα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ΑΕΠ και τη συλλογή φόρων από αυτού. φορολογική προσπάθεια. Αυτό σημαίνει πόσοι φόροι συλλέγονται σε σχέση με εκείνους που θα μπορούσαν να συλλεγούν στο σύλλογο. Έχει μειωθεί αυτό στις φτωχές χώρες την τελευταία δεκαετία. Ας πούμε, στην απόδοση ΦΠΑ ε, το διαφυγόν κέρδος είναι μέχρι και 60% της οικονομίας. Είναι τεράστιο το δυναμικό που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Τώρα, η μόχλευση των πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, είδαμε ότι πρέπει να γίνει καλύτερα και μπορεί να γίνει καλύτερα εις δίτ μπορούν να χρηματοδοτούν την υποδομή, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά όχι μόνο αυτό και διάφορα άλλα έργα υγιεινής, ανάπτυξη ακόμα και ε, του θεσμικού ε, συστήματος μια χώρα, χώρας για τη θεσμική θωράκιση. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Act Initiative. Είναι μια πρωτοβουλία για ειδικέ επενδύσεις στους τομείς που βλέπετε εδώ στη διαφάνεια που ε, καλύπτεται μόνο, πληρώνονται τα ποσά ε, βάσει αποτελέσματος με ε, ομόλογα στις χρηματαγορές με υποσχέσεις δωρητών για μελλοντική χρηματοδότηση. Ε, ας πούμε στην περίπτωση εδώ της δημόσιας υγείας για την ανοσοποίηση για εμβολιασμούς. Βεβαίω μπορούμε πάντα να χρησιμοποιούμε καλύτερα τους πόρους που έχουμε με συγκεκριμένη στόχευση και των συνταξιοδοτικών ταμείων και διαφόρων άλλων ταμείων που είναι, ε, έχουν πολλά μεγάλα χαρτοφυλάκια, πάνω από 13 εκατομμύρια πλέον δολάρια και ιδιαίτερα τα συνταξιοδοτικά ταμεία μπορούν να παίξουν ρόλο στη χρηματοδότηση τέτοιων δομών, τέτοιων προβλημάτων, υποδομών κτλ. Δηλαδή και έτσι μπορούμε να έχουμε ένα πιο έξυπνο, πιο ευφύ τρόπο χρηματοδότησης και εξέβρεση κονδυλίων για την ανάπτυξη. Μάλιστα, όλα αυτά θα γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικά αν τα κάνουμε και σε εταιρική σχέση. Ξέρουμε για την περίοδο μετά το 2015 που είναι για όλους μας προτεραιότητα, ε, χρειάζεται συντονισμός και γι' αυτό όπως και εσείς προβαίνουμε και σε συστάσεις. Να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο με στόχους, με δείκτες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμμετέχει στην ε, αντίστοιχη επιτροπή που έχει στόχο την καλύτερη υλοποίηση, εφαρμογή και έλεγχο αυτού του πλαισίου. Νομίζουμε ότι και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Συμπέρασμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει πιο αποτελεσματική η βοήθεια, να έχει ε, μόχλευση επιπλέον χρηματοδότησης και όλα αυτά από κοινού με συνεργασία. Έχω άλλες δύο διαφάνειες για το πώς μπορεί να βοηθήσει η Παγκόσμια Τράπεζα σε συνεργασία. Γενικά συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στον κόσμο με διάφορους φορείς. Εδώ βλέπετε στη διαφάνεια αυτή τι μπορούμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Ε, και για το πλαίσιο του 2015 ε, για να υποστηρίξουμε την αναπτυξιακή ατζέντα. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει και με τις στατιστικές δυνατότητες που έχει, γιατί είπαμε ότι είναι βασικό στοιχείο αυτό για την αποτελεσματικότητα ζωτική σημασία στις σωστές στατιστικές. Μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε επίπεδο κρατών, ε, έλεγχο των εθνικών στρατηγικών και ε, ανάπτυξη προγραμμάτων που να βασίζονται και να κρίνονται από το αποτέλεσμα. Και τέλος μπορούμε να συνεργαστούμε ε, για καινοτόμους μηχανισμούς όπως το blending, η ανάμειξη διαφόρων και η μόχλευση διαφόρων πηγών. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνω την παρουσίασή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Σοφή Σιρτέν και να περάσουμε στον τελευταίο ομιλητή του πρώτου πάνελ, ο κύριος Τζέσι Γκρίφιθ, διευθυντής του Eurodad, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Χρέος και την Ανάπτυξη, ο οποίος έχει ευρεία εμπειρία ε, για, στα χρηματοπιστωτικά και θα μας ε, μιλήσει για, με θέμα την βελτιστοποίηση των πόρων, των αναπτυξιακών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Συνήθως ήθιστε ε, ε, να, ήθιστε να ευχαριστεί κανείς ότι πολύ ωραία ήταν αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα και συμφωνώ, αλλά εγώ πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι ε, ευγενής και να συμφωνήσω. Θα επανέλθω όμως αργότερα σε αυτό. Ε, θέλω να πω τρία κεντρικά θέματα. Πρώτον, μιλάμε για την ανάγκη βελτιστοποίησης ε, των πόρων και την εξέβρεση νέων βελτιστοποιημένων ε, μηχανισμών. Αλλά να μην ξεχνήσουμε ότι μιλάμε για μεγάλη ανάγκη παραδοσιακών πόρων, δημοσίων πόρων. Δεύτερον, ε, το blending αυτό, καθώς επίσης και η μόχλευση των ε, ιδιωτικών κεφαλαίων ε, μπορεί να καταστεί εξαιρετικά προβληματικό. Τρίτον, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στα πλαίσια της ανάγκης να στηρίξουμε την κινητοποίηση ημεδαπών εγχωρίων πόρων. να ε, καταπολεμήσουμε τις ε, ε, χρηματοδοτικές ροές τις παράνομες και επίσης να χρησιμοποιηθούν οι σωστές διαδικασίες έτσι ώστε ε, οι μεδαπές ε, στατικές ε, να δώσουν καλά αποτελέσματα. Όσον αφορά το πρώτο μου ζήτημα, την μεγάλη ανάγκη για δημόσια, δημόσιους πόρους, είναι πολύ διαφορετικά, διαφορετικοί υπολογισμοί Εάν ε, για το 2015 και μετά θέλουμε να θέσουμε ε, πιο φιλόδοξους στόχους, τότε ε, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια στοιχεία. όσα ΣΑΑ αναφέρεται σε 60 δις για τις ιατρικές ανάγκες του κόσμου. Το Ηνωμένα Έθνη σε ένα τρεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Έχουμε 37 χώρες ε, οι οποίες είναι χαμηλού εισοδήματος ε, και προς τις οποίες ε, η βοήθεια αντιπροσωπεύει πάνω από 10% του ΑΕΠ. Το δεύτερο μου τώρα θέμα, το οποίο αφορά την μόχλευση που προκύπτει από τα ιδιωτικά τους ιδιωτικούς πόρους και τις ιδιωτικές ε, εταιρείες. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα προβληματικό το ότι έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί πρώτον έχει την τάση να ακολουθεί την αγορά ε, και επομένως ε, οι μεγαλύτερες επενδύσεις γίνονται όχι στις χαμηλές οικονομικές χώρες, αλλά στις μέσες τρία τέταρτα των επενδύσεων πηγαίνει στις μεσαίες χώρες. Επίσης, ε, ε, προωθούνται προς ε, γνωστούς κλάδους με τους οποίους έχει ήδη ασχοληθεί το χρηματοπιστωτικό πλαίσιο και όχι σε καινοτόμους όρους. Επομένως, φτάνουμε στην επόμενη ερώτηση. Ποιος κάνει τη μόχλευση? και ποιος μοχλεύει τι και ποιον, πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα πώς έχουν τα πράγματα εδώ. Ας πούμε, από την Κομισιόν έχουμε αυτόν τον αριθμό ε, του λόγου 30 προς 1 όσον αφορά την ε, μόχλευση αλλά από εδώ προκύπτουν και από αυτό το αριθμητικό στοιχείο προκύπτουν ε, πολλά ε, ερωτήματα, δηλαδή τι συμβαίνει, τι μπορεί να συμβεί, ε, τι γίνεται με αυτούς τους ιδιώτες επενδυτές που ούτως ή άλλως θα επένδυαν. Επίσης, εάν ε, ο λόγος μόχλευσης ξεπεράσει και το 30 προς 1, γιατί εγώ έχω ακούσει και κάτι τρομερά στοιχεία, 100 προς 1, ε, τότε πού φτάνουμε και προς τα πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά, με ποιο τρόπο δαπανώνται, σε τι προγράμματα δαπανώνται. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Και προκύπτει και κάτι άλλο. Υπάρχει τεράστιο κόστος ευκαιρίας. Ε, ξέρουμε ότι κάθε δολάριο το οποίο ε, ξοδεύουμε ε, και το βάζουμε στη μόχλευση είναι ένα δολάριο το οποίο αφαιρούμε από τις παραδοσιακές, από τους παραδοσιακούς τρόπους επένδυσης και βοήθειας. Επομένως, ε, πρέπει να μας προβληματίζει πάρα πολύ αυτή η πολύ ασθενής λογοδοσία και διαφάνεια. Κοιτάξτε, ε, ο διαμεσολαβητής, ο Ombudsman για την ε, Παγκόσμια Τράπεζα έχει αναφερθεί σε όλα αυτά τα προβλήματα ε, και συμπερασματικά πάντως είπαν ότι η Παγκόσμια Τράπεζα δεν ήταν σε θέση να ελέγξει το περιβάλλον αυτών των επενδύσεων, τουλάχιστον στις περισσότερες από τις περιπτώσεις και, και στα περισσότερα χαρτοφυλάκια ξέροντας ε, τι συγκίνεται με τα χρήματα, ξέροντας την ελληπή λογοδοσία, την ελληπή ε, διαφάνεια, προφανώς ε, προβληματιζόμαστε ιδιαίτερος. Και βεβαίω βεβαίως προκύπτει και το τελευταίο ερώτημα το οποίο μας απασχολεί πολύ. Αν τα πράγματα πάνε άσχημα, ποιος θα πληρώσει, ε, ποιος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει το ρίσκο του ε, χρέους, και όταν ε, ακούω δεξιά-αριστερά να λέγεται ότι πρέπει η μόχλευση στι αναπτυσσόμενε χώρε να είναι μεγαλύτερη, εγώ λέω για σταθείτε μια στιγμή, πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. ποια είναι η εναλλακτική λύση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους αναπτυξιακούς πόρους έτσι ώστε να στηρίξουμε την κινητοποίηση των εγχωρίων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν στα τέλη του προηγούμενου έτους εμείς κάναμε ένα κατάλογο όλων των βαθμίδων. Ε, σε, με μπλε χρώμα βλέπετε τις, ε, τους εγχώριους πόρους που κατά πολύ ξεπερνούν τους ε, άλλους χώρους. 20% του ΑΕΠ ενώ και υψηλό είναι και το ποσοστό της ιδιωτικής επένδυσης. και εάν δει κανείς προσεκτικά και τους κόκκινους ε, αριθμούς, ε, τότε βλέπετε ότι ε, αυξάνονται και ο κυβερνητικός δανεισμός αλλά και οι παράνομες ροές, ενώ δηλαδή εγκληματικές έγκλημα, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή κτλ. Ε, και νομίζω ότι σε όσους βουλευτές είναι παρόντες θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή τους ε, σε αυτή την οδηγία για το ξέπλυμα ε, μαύρου χρήματος. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει εδώ να αναφέρω είναι το πώς χρησιμοποιούμε τα χρήματα όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Περίπου το μισό του συνόλου της βοήθειας επενδύεται μέσω του ιδιωτικού τομέα. Δύο τρίτα αυτής της βοήθειας πηγαίνει σε εταιρείε των χωρών ΩΣΑ. Στην ουσία δηλαδή διοχετεύουμε την ε, αναπτυξιακή ε, βοήθεια και την ε, ανακυκλώνουμε. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα με μια διαφορετική κατανομή χωρών. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να προωθήσουμε τα πράγματα. Αλλά βλέπετε ότι μέχρι τώρα ε, υπάρχουν πολλές ε, ε, χώρες στις οποίες υπάρχει μία anti-aid συμφωνία. όπου δεν είναι δυνατόν να επενδυθεί το 60% της αναπτυξιακής βοήθειας μέσα από δημόσιους φορείς. Λοιπόν, να μην λησμονούμε εν συμπεράσματο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη από παραδοσιακές ε, δημόσιες χρηματοδοτήσεις. Δεύτερον, ε, να μην μπερδεύουμε πολύ τα πράγματα γιατί το blending και η υπερβολική μόχλευση οδηγούν σε επιπλέον ε, προβλήματα Τρίτον, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα στην κινητοποίηση των εγχωρίων πόρων να, με τρόπο ώστε να αποφύγουμε τις παράνομες εκροές χρημάτων να καταπολεμήσουμε ε, προβλήματα όπως είναι το, ε, το ξέπλυμα χρήματος και η φοροαποφυγή ε, και να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα επιθυμούσαμε. Πάρα πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το πρώτο πάνελ και περάμε στο δεύτερο πάνελ, στη δεύτερη ομάδα ε, εκεί θα έχουμε εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μας δώσουν συγκεκριμένα γεωγραφικά παραδείγματα πραγματογνωμοσύνης και επιτυχημένων προσπαθειών. Ο κύριος Ντέρκ Βίλεμ Τεβέλντε είναι ο, ο πρώτος, ο οποίος θα πάρει την, την το λόγο. Είναι επικεφαλής ομάδας Διεθνούς Οικονομίας και ανάπτυξη του Υπερπόντιας Ανάπτυξης Overseas Development Institute. Είναι μέλος ε, της ε, ομάδας ε, της Think Tank για το blending του 2011 με μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε δωρητές και διεθνείς οργανισμούς. Ο κύριος Τεβέλντε θα μας δώσει μια κριτική επισκόπηση ε, για τις διευκολύνσεις blending της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Ντεβέλτε μου, έχετε το λόγο. Α, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας από το εκ μέρους του ODI. Ήδη έγινε μια πρώτη εισήγηση κυρία Πρόεδρε και ξέρετε ότι και εμείς έχουμε μελετήσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα blending. Τρία πράγματα θέλω να κάνω. Πρώτον, να σας περιγράψω το blending γενικότερα, το πλαίσιο του μάλλον. Στην αρχή σκεφτόμασταν την αναπτυξιακή βοήθεια που ήταν η μόνη χρηματική πηγή για την ανάπτυξη για ορισμένες χώρες, ενώ τώρα μιλάμε για διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Είχα σχεδιάσει να μιλήσω λεπτομεριακά για τις ε, δυνατότητες blending στην Ευρώπη, αλλά Χωσέ, ο Χωσέ τα περιέγραψε καλά και μπορώ εκεί να τα παραλείψω. Και μετά θα καταλήξω για τα υπέρ και τα κατά των προγραμμάτων blending με βάση μελέτες μας από συγκεκριμένα προγράμματα blending και από μελέτες από διάφορες δεξαμενές σκέψεις. Λοιπόν, πρώτα, Ας δούμε πώς έχουν γενικότερα τα πράγματα με τη χρηματοδότηση ή τη χρηματοπίστωση. Οι προηγούμενοι ομιλητές είπαν μερικά για την κινητοποίηση εγχωρίων πόρων, πολύ σημαντικός πόρος και αυτός. Ταυτόχρονα όμως υπά... σημειώθηκαν αλλαγές και σε αυτό. Παραδείγματο χάρη στην Υποσαχάρη Αφρική έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι χρηματοδοτήσεις και δεν μιλάμε μόνο για εξωτερικές επενδύσεις αλλά και για άλλε μορφές ομολόγων α πούμε και κίνησης ομολόγων. Πολλές χώρες στην Αφρική αυτή τη στιγμή έχουν ε, δημιουργήσει ομόλογα χρεώνονται δηλαδή περισσότερο και υπάρχουν και άλλες χρηματοπιστωτικές ροές Aid for Trade, ODA και άλλα. Βασικά λοιπόν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάφορες μορφές χρηματοδοτικών ροών. Το blending συνδυάζει δωρεές και δάνεια. Δάνεια βέβαια σημαίνει και χρέωση της χώρας που τα παίρνει. Στην υποσαχάρη Αφρική ας πούμε βλέπουμε ότι το χρέος ήταν για πολύ καιρό σταθερό και μετά αυξήθηκε απότομα. Και από την άλλη Μειώθηκαν οι εξαγωγές, ίσως, οι εισαγωγές μάλλον, λόγω της βοήθειας ίσως. Σε άλλες χώρες έχει σταθεροποιηθεί, δηλαδή σταμάτησε η μείωση. Επίσης πιστεύω ότι οι χώρες που δέχονται τέτοιου είδους χρηματοδότηση συνεχώς ζητούν και περισσότεροι, δέχονται την αύξηση του χρέους τους δηλαδή παραπάνω από ό,τι μπορεί να τους δώσει η απλή ανθρωπιστική βοήθεια. Ένα πρόσφατο παράδειγμα που συζητήσαμε πρόσφατα ήταν η Ρουάντα. Ομόλογα 400 εκατομμυρίων. Σε εποχή μάλιστα που μειώνονταν η βοήθεια. Όλο και περισσότερο λοιπόν οι χώρες που παίρνουν τέτοια χρηματοδότηση θεωρούν ως δέσμη, συνδυασμό όλες αυτούς τους τύπους ροών. Οδικές υποδομές και άλλα πρέπει να χρηματοδοτηθούν και αναρωτιούνται πώς να το πετύχουν καλύτερα με εξωτερικές επενδύσεις, με δωρεές, με δάνεια. Θέλουν όμως πάντως να γίνει η επένδυση για να υπάρξει περισσότερη ανάπτυξη είτε στις υποδομές είτε στην ενέργεια και αν υπάρξει ανάπτυξη θα αυξηθούν οι πόροι και οι χώροι για να αντιμετωπιστεί η ανέχεια και να βελτιωθεί η υγειονομική περίθαλψη. Βασικά λοιπόν οι χώρες αυτές επιζητούν δέσμες, blending δηλαδή, Όλα αυτά βέβαια γίνονται σε θεσμικά πλαίσια όπου παίζουν πολλοί παράγοντες. Υπάρχουν πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ευρωπαϊκά και μη, διάφορων ειδών τράπεζες όπως η τράπεζα των λεγόμενων BRICS, φιλανθρωπικές οργανώσεις, επενδυτές κλπ. Είναι δύσκολο λοιπόν να καθορίσουμε ακριβώς ποια θέση θα να παίξει η Ένωση σε αυτά. Κάτι που μπορεί σίγουρα να κάνει είναι να συνδυάσει τους πόρους που διαθέτει. Και ορισμένες μεμονωμένες χώρες συνδυάζουν τους πόρους που διαθέτουν όπως έγινε στη Γαλλία. Και σε ενωσιακό επίπεδο θα μπορούσαν να συνδυαστούν όλα αυτά πιο αποτελεσματικά. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά για τα προγράμματα blending τα ίδια γιατί έγινε η παρουσίαση από την Κομισιόν. Θα ήθελα απλώ να πω ότι οι δωρεές χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους. Ένας από τους απλούστερους είναι ότι μπορεί να χρηματοδοτήσουν μία μελέτη αξιολόγησης ή κόστους οφέλους που χρειάζονται για να γίνει μια επένδυση. Αν δεν έχουν γίνει αυτές οι μελέτες δεν θα αναλυφθεί το σχέδιο, κανένα σχέδιο. Μερικά και τέτοιε μελέτες βέβαια χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν και πολύ τεχνική βοήθεια. Κάποιος πρέπει να τις χρηματοδοτήσει και να αναλάβει τον κίνδυνο. Σε μερικές από αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν το αποφασιστικό βήμα είναι ποιος θα χρηματοδοτήσει την έγκριση, την προκαταρκτική έγκριση αυτών των σχεδίων. Θα ακούσατε πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τη βοήθεια που χορηγείται σε προγράμματα blending και το ρυθμό της μόχλευσης, την αναλογία της μόχλευσης, τον λόγο της μόχλευσης. Η τελευταία μου διαφάνεια θα μιλήσει για τα υπέρ και τα κατά. Τα υπέρ του blending είναι ότι βοηθάει να απελευθερωθούν χρηματοδοτήσεις. Όπως σας είπα πριν παραδείγματο χάρη χρηματοδότηση μίας μελέτης κόστους ωφέλους ή αξιολογήσεις. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει η χρηματοδότηση και μελέτη για επενδύσεις είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, το είπαν και άλλοι. Αν δείτε ποιος είναι ο κύριος φραγμός στην ε, ανάπτυξη, δε, συνήθως δεν είναι οι υποδομές και οι μεταφορές, αλλά είναι μάλλον οι υποδομές και οι μεταφορές και εδώ μπορούν να βοηθήσουν τα προγράμματα blending. Μετά είναι οι εντυπωσιακοί λόγοι μόχλε, της μόχλευσης και μετά η ευελιξία των λύσεων αυτών. Δεν μπορεί κανένας μεμονωμένος οργανισμός να χρηματοδοτήσει ολόκληρο δρόμο από δωρεές ή έναν υδροηλεκτρικό ή άλλο σταθμό. Χρειάζονται μαζικά ποσά και γι' αυτό χρειάζεται ολόκληρη δέσμη πόρων. Και βέβαια η, το blending έχει οδηγήσει και σε καλύτερο συντονισμό και ορατότητα. Επίσης η Κομισιόν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα για καλύτερο συντονισμό για την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων. Πολύ καλό πράγμα αυτό. Τώρα ορισμένες προκλήσεις ή αρνητικά σημεία. Πρώτον, ο ορισμός. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό αυτά τα νέα προγράμματα blending μπορούν να θεωρηθούν σαν αναπτυξιακή βοήθεια. Το θέμα είναι αν καταμετρούνται όλα τα συστατικά ενός προγράμματος blending. Ίσως μόνο ένα τμήμα τους να μπορεί να θεωρηθεί σαν αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά εμείς μετράμε τη γενική επίπτωση μιας δέσμης, αν καταλήγει σε ανάπτυξη ή όχι. Πρέπει πρέπει προηγουμένως να έχουμε ορίσει έναν σφαιρικό γενικότερο αναπτυξιακό στόχο για να τα κρίνουμε όλα αυτά. Τώρα κάτι πιο ουσιαστικό, οι λόγοι μόχλευσης. Τζέσι και ο Χωσέ είπαν μερικά αλλά ε, η δική μου θέση είναι ανάμεσα στους δύο. Λόγος 1 προς 30 μπορεί να μην σημαίνει κάτι το αντικειμενικά βέλτιστο. Είναι εξαρτώνται όλα αυτά από τους στόχους. Εμείς κάναμε μια ανάλυση της λειτουργίας των αναπτυξιακών ιδρυμάτων ιδίω ιδιωτικά και διαπιστώσαμε το εξής, αναρωτηθήκαμε μάλλον το εξής ποια είναι ποιο είναι το όφελος από όλα αυτά ένα προς τέσσερα, ένα προς πέντε, ένα προς τριάντα είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα και πώς. Κάναμε λοιπόν μια μελέτη που εξέταζε τις επενδύσεις από τη μία και τα αποτελέσματά τους από την άλλη και τα συγκρίναμε με το ΑΕΠ και, άλλους, και άλλα κριτήρια που συνήθως λαμβάνονται υπόψη στις επενδύσεις για να δούμε αν οι αναπτυξιακοί πιστοτικοί οργανισμοί δουλεύουν. Βρίσκουμε εδώ μερικά θετικά στοιχεία και συμπαράσματα, όχι όμως παντού ούτε πάντα. Αυτό θα μπορούσε κανείς να το περιμένει. Υπάρχει μια σειρά αποτελεσμάτων από διαφορετικά πιστοτικά ιδρύματα με διαφορετικά αποτελέσματα. Σε μερικά η μόχλευση και μόνο ένα προς δύο είναι αποτελεσματική. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, όχι. Χρειάζονται βέβαια περισσότερες μελέτες εδώ, αλλά βλέπουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις είναι καταλητικά τα αποτελέσματα του λόγου και σε άλλα όχι. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε λοιπόν, να δούμε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει στο blending. Εδώ συμφωνώ με τον Τζέσι λοιπόν. Τον Τζέσι, τον Ιεσέ. Και τώρα η διακυβέρνηση. Αυτό το προσέξαμε ιδιαίτερα και υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία λέει ότι η αναπτυξιακή στόχη είναι το κυριότερο ενώ η άλλη το κατά πόσον υπάρχει ιδιωτικός τομέας ή μια εταιρεία του ιδιωτικού τομέα που συμμετέχει στη χρηματοδότηση και μπορεί να αναλάβει τον κίνδυνο και θέλει να επενδύσει. Αλλά όλα αυτά πρέπει να είναι βιώσιμα, δηλαδή να αποφέρουν κέρδη. Πάντως υπάρχουν δύο τρόποι να το δει Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις, μάλλον σχέδια, έχουν καλύτερα αποτελέσματα και στην οικονομία γενικότερα, αλλά όχι απαραίτητο. Και άρα το ερώτημα τίθεται ποιο είναι το κυριότερο στοιχείο, Ποιες προτάσεις ε, μιας δέσμης με ενός προγράμματος είναι οι πιο αποτελεσματικές και πώς να κρίνει κανείς αν είναι καθοριστική η πλευρά της αγοράς ή όχι ή των δωρεών. Δεύτερον, μήπως χρειάζεται, χρειάζονται περιφερειακά προγράμματα blending ή θεματικά ή μήπως να συνδυαστούν. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά για κάθε περίπτωση και για τις τρεις αυτές περιπτώσεις. Πώς θα διασφαλίσουμε όμως πώς οι πόροι να πάνε σε ποιο θέμα και σε ποια περιφέρεια. Και βέβαια ποιες χώρες να αφορά. Ποιες χώρες να πάρουν τι. Δεν έχουν ώρες όλες τον ίδιο ρυθμό δανειοληψίας ή δανειοληπτικής ικανότητας. Τι εργαλεία διαθέτουμε για να τα καθορίσουμε ή να τα κρίνουμε όλα αυτά. Εδώ χρειάζεται περισσότερη ανάλυση για να το βρούμε μέσω στη διακυβέρνηση βέβαια. Τέλος, τέλος λέγω, ποια είναι η σύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα. Η πρώτη παρουσίαση είχε πει ότι τα θε... blending αφορά κυρίως τον δημόσιο τομέα. Πριν από δύο χρόνια όταν τα εξετάζαμε τέτοια σχέδια ήταν σχεδόν όλα από το δημόσιο τομέα. Δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να αποκλείσουμε βοήθεια και από και για τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα βοηθούσε πάρα πολύ να γίνει η ανάπτυξη από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί οι παραγωγικές επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερη απασχόληση και περισσότερη κινητοποίηση εγχωρίων πόρων. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα θέμα του πώς να συνδυαστούν όλα αυτά με τον ιδιωτικό τομέα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm. Καταλήγω λοιπόν ότι πρόκειται για ένα νέο τρόπο εδώ, το blending δηλαδή, συνδυασμού διαφόρων πόρων, είναι όμως ο δρόμος του μέλλοντος. είτε πρόκειται για τις χώρες BRICS, είτε για την Κίνα, είτε για το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλους. Είναι πολύ χρήσιμος τρόπος συνδυασμού πόρων, αλλά πρέπει να δούμε κάτι παραπάνω για τη διακυβέρνηση, για τα εργαλεία που διασφαλίζουν ότι οι πόροι που θα διατεθούν είναι, έχουν όντως προσθετικό χαρακτήρα και θετικές επιπτώσεις και μετά να γίνει και ανάλυση ανατομέα και αναχώρα κλπ. Σας κατευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ για την ακρίβεια της παρουσίασής σας και τώρα ερχόμαστε στην πρώτη μελέτη συγκεκριμένου παραδείγματος που έχει να κάνει ε, με τη συνεργασία με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με ζητήματα χωρών σε προταξιακό καθεστώς στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ομιλητές μας. Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο κύριος Καράνο και ο κύριος Τσιγκολάνη, αν διαβάζω καλά το όνομα σας. Ο Αλεσάνδρο Καράνο ε, είναι σύμβουλος διευθυντικός και τμήματάρχης ε, στο τμήμα ε, θεσμικής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και συνεισέφερε στη πλατφόρμα για το blending στο πλαίσιο επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια και άλλους τέτοιους μηχανισμούς. Ο Μάσιμο Τσιγκολάνη ε, είναι επίσης σύμβουλος και ε, αναπληρωτής τμήματάρχης ε, στο τμήμα Αδριατικής και συντονίζει θέματα Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο και που καλέσατε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μιλήσει στην τόσο ενδιαφέρουσα αυτή ακρόαση. Εγώ θα μιλήσω για 10 λεπτά και ο συνάδελφό μου ε, θα απαντήσει στις δύσκολε ερωτήσει που θα το κάνετε. Δηλαδή μισό-μισό θα το μοιραστούμε το χρόνο μα. Καταρχά θα ήθελα να σα πω ποια είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων απέναντι στο blending ε, ε, και ιδιαίτερα τη δημιουργία του πλαισίου επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Μάσιμο Τσιγκολάνη θα σα δώσει κάποια πρακτικά παραδείγματα στη συνέχεια, καθώ επίση και ε, την εμπειρία ε, με τα έργα που έχουμε σε αυτό το πλαίσιο. Και ε, κάποια αντίστοιχα για το μέλλον που προβλέπουμε. Πολύ σύντομη εισαγωγή. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπω γνωρίζετε, χρηματοδοτεί κυρίω έργα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υποστηρίζουμε και τις εξωτερικές πολιτικές, κυρίω τη διεύρυνση και τη συνεργασία με χώρες ε, για την ανάπτυξη και για το κλίμα και το περιβάλλον, ε, όπως έχει ε, καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες εκτός της Ένωσης επαναλαμβάνω και αυτό είναι περίπου το 10% των ετησίων μας δραστηριοτήτων. 7 δις ετησίως με blending πάλι προς χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, για το δημόσιο αλλά και για το ιδιωτικό τομέα, τα έργα δηλαδή. Ε, έχουμε εντολή που συμπίπτει με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικό αυτό όμως, προσέξτε γιατί. Είναι και ένα μέσον που επιτρέπει να συνδυάζουμε διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Γι' αυτό ε, βασίζεται και σε μια ε, ε, εγγύηση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι μπορούμε να καλύπτουμε και τον πολιτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο για τα κράτη. Ε, που είναι εγγενής ε, ε, για την τράπεζά μας για δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούμε έτσι να χορηγούμε δάνεια με τα χρήματα που αντλούμε από τη χρήματα αγορά. Στο παρόν χρηματοδοτικό πλαίσιο, το πολιετές, μέχρι τέλη του έτους έχουμε 30 δις blending με δάνεια με εγγύηση από τον προϋπολογισμό κόμμα 12 δισεκατομμύρια στον προπολογισμό. Από πηγέ ε, είπαμε, δανειζόμαστε από τις χρηματαγορέ για να χορηγήσουμε τα δάνεια στη συνέχεια. Ε, η πρόταση πρόσφατα πέρασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, είναι θέμα συναπόφαση του, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου προσεχώς ε, προσβλέπουμε σε αυτή την έγκριση της ε, εντολής μας, γιατί δεν είναι μόνο εγγύηση, αλλά θέτει και το πλαίσιο της πολιτικής και όλες τις απαιτήσεις για το blending, για τη δημιουργία της πλατφόρμας και άλλες απαιτήσεις για την αναπτυξιακή επίπτωση των δραστηριοτήτων μας. Όλα αυτά απορρέουν από ε, εκείνους που χαράσουν την πολιτική και μάλιστα είναι και κείμενα με νομική αξία αυτά και ισχύ. Ιδιαίτερα λοιπόν για το μείγμα αυτό του blending έχουμε αναπτύξει δραστηριότητες, συνεργασία και εμπειρία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δεν θέλω καθόλου να επαναλάβω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες Συμφωνώ με μερικά σχόλια για τη μόχλευση πάντως που είναι πολύ σημαντική ως έννοια από μόνη της. Ταυτόχρονα όμως θέλει λίγη προσοχή για τους αριθμούς που παραθέτουμε διότι είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε ε, δωρεές για τεχνική βοήθεια, για μελέτη σκοπιμότητας ή ε, για επενδύσεις ή άλλου τύπου δωρεές. Δεν είναι η ίδια η μόχλευση ούτε η ερμηνεία ανάλογα με το έργο και επίσης το blending δεν είναι, ένα blender δεν είναι ένα μηχάνημα που κόβει λεφτά, αλλά δημιουργεί με τη μόχλευση και με το συνδυασμό προστιθέμενη αξία λόγω της πραγματογνωμοσύνης και όχι μόνο των χρηματών και των πηγών χρηματοδότησης και των πόρων. Για να ε, Έχουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς το στόχο που έχει χαρακτεί κάθε φορά. Αναφέρθηκε η ποιότητα των προγραμμάτων, ε, η αηφορία τους και η βιωσιμότητά τους, αλλά έχουμε και πάρα πολύ σαφείς προδιαγραφές όταν δίνουμε ένα δάνειο, το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί μετά από μια σειρά ετών. Και παίρνουμε τις προφυλάξεις μας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κρατικές προμήθειες, αλλά ε, και περιβαλλοντικά στοιχεία και πρότυπα άλλα συμμόρφωσης ε, που είναι ουσιαστικά ε, ιδέουσα επιμέλεια στην ουσία της. Κάτι άλλο που έχει να κάνει με τα δάνεια επίσης πολύ σημαντικό και επιτρέπει στο δικαιούχο να κάνει κτήμα του αυτό το σύστημα είναι ο τρόπος αποπληρωμής ε, με την πάροδο του χρόνου. Επανειλημμένα ε, ακούσαμε για συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων εταίρων. Να σας δώσουμε μερικά παραδείγματα. Ε, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η BERD λοιπόν και οι τράπεζά μας μπορούν να έχουν κοινά έργα και κοινέ δραστηριότητε σε όλες τις χώρε γειτονία και τις προενταξιακέ. Ε, και από πολύ νωρί να σχεδιάζουμε κοινά έργα και δράσεις όπου χρειάζεται φέρει πίνση χρηματοδότηση. Ε, και έχει τριπλασιαστεί η χρηματοδότηση το τελευταίο διάστημα από τότε που δημιουργήθηκε το ε, μέσον αυτό. Τα μισά από τα ε, προγράμματά μας εκτός Ένωσης είναι συγχρηματοδοτούμενα με άλλες τράπεζες, άλλα πιστοτικά ιδρύματα, είτε είναι αυτά ευρωπαϊκά είτε διεθνή. Άλλο παράδειγμα, ε, η πρωτοβουλία αμοιβαίας ανάληψης και ε, στην Αφρική και στην Υποσαχάρη έτσι ώστε πολύ νωρίς εντοπίζουμε τα προγράμματα της δραστηριότητές μας για να ξέρουμε ποιο θεσμός, ποιο ίδρυμα είναι σε καλύτερη θέση για να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο ε, για ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να έχουμε ένα πιο ορθολογικό επιμερισμό ε, της εργασίας παρά να έχουμε παράλληλη ναι, ναι. και επικάλυψη στη δράση μας. Έχουμε λοιπόν διαδικασίες για τα δάνεια ε, και με τη δέουσα επιμέλεια ακριβώς ακολουθούν και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να μην υπάρχουν διπλές δουλειές και επικαλύψεις και παράλληλες προσπάθειες. Ακούσαμε και προηγουμένως τοποθέτηση Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά. Έρχομαι τώρα στο ειδικό παράδειγμα ε, του πλαισίου επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και χαιρόμαστε πολύ αυτό γιατί μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, τα κράτη-μέλη και άλλα τεινά, το 2009 το ρυθμίσαμε το πλαίσιο αυτό. Δεν ήταν εύκολη προσπάθεια, ούτε απλή, γιατί έπρεπε να καθοριστούν ε, διάφορα στοιχεία του μηχανισμού αυτού για τη διακυβέρνηση, όπως υπόθηκε και προηγουμένως. Ένα από τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να προσέχουμε είναι αυτό, έτσι ώστε να ε, παντρεύουμε τις ανάγκες και τις ανησυχίες των δωρητών με των δικαιούχων. Ε, χρειάστηκε λίγος χρόνος λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που καταφέραμε να το λασάρουμε τότε και στη συνέχεια να το βελτιώσουμε λίγο για να μπορούμε να συνενώνουμε τους πόρους των δανείων ή των, των δωρεών ε, σε ένα πλαίσιο γιατί στο παρελθόν ήταν κατακαιρματισμένα. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έδινε χρήματα ορισμένα κράτη-μέλη με δικά τους ταμεία, ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλες παράλληλες χρηματοδοτήσεις είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους δωρητές. Εδώ λοιπόν καταφέραμε να συνενώσουμε όλα αυτά τα μέσα σε ένα πλαίσιο, πράγμα το οποίο εκτίμησαν σφόδρα οι ε, δικαιούχοι αλλά και τα κράτη-μέλη μας και μπορούν τα κράτη να δίνουν δωρεές έτσι που δεν μπορούσαν στο παρελθόν να χορηγούν ε, στις περιφέρειες, αλλά το έκανα μόνο σε διμερή βάση. Λοιπόν, μία είναι η ε, δραστηριότητα λοιπόν για τις προτεραιότητες ε, στην πολιτική διεύρυνση, τα ορίζουν αυτά μόνοι τους οι ε, δικαιούχοι, αποδέκτες, μας ζητούν δηλαδή ακριβώς τι θέλουν και βεβαίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη συνέχεια εξετάζουν τα αιτήματα και αποφασίζουν ανάλογα με τις δυνατότητες ε, χρηματοδότησης. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο καταφέραμε να δίνουμε και πόρους από τους ιδίους πόρους μας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να μεγιστοποιήσουμε και πάλι τη μόχλευση, διότι δεν δίνουμε μόνο δάνεια, αλλά τα τρία χρηματοδοτικά ε, χρηματοπιστωτικά Ινστιτούτα δίνουν και χρήματα από το προπολογισμό. Αφήνω να το λόγο τώρα στο Μάξιμο Τσιμπολάν. Ευχαριστώ πολύ, Αλεσάνδρο. Θα συνεχίσω λέγοντας ότι πολύ σωστά αναφέρθηκες σε αυτόν τον συντονισμό της ε, βοήθειας ε, μέσα σε αυτόν τον μηχανισμό ανάμειξης. Ενδιαφέρον είναι να δει κανεί ε, ότι στην αρχή ναι, το αίτημα για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των δωρητών έχει προέλθει από την από το αίτημα των ε, ιδίων των ε, βοηθουμένων. Ε, δηλαδή ζήτησαν από τους δωρητές να συνεργαστούν μεταξύ τους, έτσι ώστε και η εφαρμογή και η υλοποίηση των προγραμμάτων να είναι πιο σωστή. Επίσης και σε σχέση με αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακούσαμε μέχρι τώρα, η ιδέα αυτού του πλαισίου επένδυσης ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια ε, βεβαίως βασίστηκε ε, στα, στις και τα δάνεια, αλλά στην ουσία αυτό σημαίνει διασύνδεση μεταξύ των προγραμμάτων και της χρηματοδότησης. Δηλαδή, ταμιακή χρηματοδότηση από τη μία και project από την άλλη. Με χρήση ε, πολλών πόρων και πολλών δυνατοτήτων που αν υλοποιηθούν σωστά την κατάλληλη στιγμή ε, καταρχήν θα είναι σε θέση να γεννήσει ε, εισόδημα στο μέλλον. Και εδώ έχουμε λοιπόν έναν πραγματιστικό, μια πραγματιστική διασύνδεση. Τώρα, με ποιο τρόπο υλοποιείται αυτό το blending στα πλαίσια του ε, πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, όπως ε, είπε και ο συνάδελφος πριν εδώ, απορρέει όλη αυτή η συζήτηση από, την, από τον κανονισμό ΕΙΠΑ και ο, τελευταίο, ο τελευταίος δικαιούχος που είναι το NIPAC προκειμένου, δηλαδή ο, ο, ένα γραφείο το οποίο ασχολείται με την ε, διευθέτηση του ΙΠΑ. Ε, υπάρχει το Project Financiers Group, ε, στο οποίο, δηλαδή είναι το PFG, στο οποίο ε, δημιουργούν, ε, στο οποίο δημιουργείται μια επιτροπή ε, η οποία ελέγχει πρώτον κατά πόσο συμμορφούνται το, το αίτημα με την πολιτική της Κομισιόν και επίσης το PFG δίνει μια κρίση, κάνει μια κρίση για το κάθε πρόγραμμα, εάν δηλαδή πρέπει να στηριχτεί ή όχι τέλος η ολοκλήρωση της μελέτης, μάλλον η έκβαση, το αποτέλεσμα της μελέτης του Project Financiers ε, Group υποβάλλεται στην Steering Committee η οποία τελικά παίρνει την απόφαση για το κατά πόσον θα υπάρξει στήριξη ή όχι και ε, ε, η υλοποίηση της επιδότησης και του δανείου γίνεται από το IFI. Για να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία, μέχρι το τέλος του 2009 είχαμε 279 εκατομμύρια σε ε, δάνεια, τα οποία δόθηκαν άμεσα σε 137 projects. projects τα οποία ε, ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί και με 2,3 ε, δις ε, εκατομμύρια δανείων που έχουν ήδη υπογραφεί από το IFI. Μπορώ να σας δώσω τώρα το αριθμητικό στοιχείο, το ποσό για τα ποσά τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί μέχρι τώρα είναι 7,7 ε, δις ε, και φτάνουν τα projects μέχρι το 2022. Το πρέπει λοιπόν να είναι κανείς ε, προσεκτικός και ακριβής, αλλά βεβαίως το σημαντικό είναι τα υπογεγραμμένα δάνεια, γιατί αυτά αποτελούν συγκεκριμένη δέσμευση και για αυτά τα ε, δάνεια ε, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει δώσει σημαντική συμβολή. Όσον αφορά την μόχλευση, Βεβαίως ε, ε, η σημαντικό είναι να υπάρξει διαφοροποίηση μεταξύ του financial και του ε, ποιοτικού, του, financial, του, του, της χρηματοδοτικής μόχλευσης και της ποιοτικής μόχλευσης και βεβαίως πρέπει να την υπόψη είναι όλοι οι δονητές, οι δωρητές μεταξύ των οποίων και το IFI. Και βεβαίως με τον τρόπο αυτό δίνεται προστιθέμενη, σημαντική προστιθέμενη αξία. Για να σας ε, δώσω κάποια παραδείγματα, ε, σας έχουμε μοιράσει και ένα μικρό έγγραφο όπου απεικονίζονται διάφορα προγράμματα. Θα μπορούσα απλώς να πω δύο λόγια παραπάνω όσον αφορά το πρώτο ε, ε, πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα έρευνας ε, στην Σερβία όπου είχαμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων μαζί με την IPA και την Κεντρική Τράπεζα για να ε, προωθηθεί ένα πρόγραμμα στην, ε, στο Βελιγράδι αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ποτέ δεν θα είχε ολοκληρωθεί ε, διαφορετικά γιατί το πρόγραμμα είχε μπλοκαριστεί λόγω έλλειψης πόρων. Επίσης έχουμε στην Αλβανία ε, δρόμους στην Ήπεθρο που έχουν οικοδομηθεί διότι η BERD μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, Επενδύσεων έχουν συνεργαστεί, έδωσαν 30% των συνολικών δανείων για την αποκατάσταση ε, των πιο φτωχών ε, περιοχών της υπαίθρου της Αλβανίας. Ε, πρόκειται για δύο παραδείγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα και δείχνουν και την ευελιξία των προγραμμάτων και ε, βοηθούνται και από το εργαλείο αυτό ε, της διευκόλυνσης του επιχειρήν ε, και το, της δημιουργίας υποδομών στο, στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι το EDIF. Το εργαλείο αυτό θέλει να βελτιώσει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ε, στην χρηματοδότηση. Υπάρχουν τέσσερις πυλώνες, δύο equity funds, ένα ε, ε, fund για τις αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένα εργαλείο εγγύησης. Με τον τρόπο αυτό έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση εταιρείε οι οποίες διαφορετικά δεν θα ήταν σε θέση να αντλήσουν κεφάλαια από τους παραδοσιακούς τρόπους. 142 εκατομμύρια ευρώ δίνονται ε, για αυτό το καινοτόμο εργαλείο για την ε, πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση. Και υπάρχει και βεβαίως ε, και το πακέτο για την καινοτομία και για την έρευνα που, που τώρα έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί αργότερα τι έχουμε μάθει από αυτό το εργαλείο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, υπογραμμίσουμε την, ε, ε, την ιδιοκτησία και βεβαίως το γεγονός ότι οι δωρητές μαζί με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητούν. Το blending διασφαλίζει το ότι το ότι τα ποσά των επιδοτήσεων ή των δανείων τελικά ε, θα προχωρήσουν και θα υλοποιηθεί ένα συγκεκριμένο project. Επίσης ε, υπάρχει η δυνατότητα ε, να προστρέξει κανείς στην τεχνική βοήθεια που σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές υπογράμμισαν με το blending αυτό δημιουργούνται πολλά, ε, δημιουργείται ένα θετικό περιβάλλον όπου τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όλων των εμπλεκομένων μπορούν να έχουν ένα καθαρό πολλαπλασιαστικό θετικό αποτέλεσμα. Πολλή συζήτηση επίσης, ε, μεγάλη συζήτηση γίνεται στην οποία συζητούν όλοι και οι δωρητές και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φωνείς. Τώρα τι γίνεται με το μέλλον και εγώ αναφέρομαι μονάχα στα Δυτικά Βαλκάνια εδώ. Εμείς ξεκινούμε από μια κατάσταση όπου ε, οι προοπτικές για τα Δυτικά ε, Βαλκάνια προβλέπεται ε, μείον 0,8% ανάπτυξη του ΑΕΠ. Άρα είναι δύσκολη η κατάσταση. Γνωρίζομαι κάνοντας κάποιους υπολογισμούς και θα σας πω δύο λόγια για αυτά στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, 14-20, θα χρειαστούμε περίπου 8 με 9 δις ε, εκατομμύρια κάθε χρόνο ε, για να επενδυθούν σε υποδομές και άλλες προτεραιότητες οικονομικής και κοινωνικής φύσεως στα Δυτικά Βαλκάνια. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσει αυτή η ιδέα του blending, γιατί ε, και οι επιδοτήσεις και τα δάνεια θα πρέπει να προωθούνται και να επικεντρώνονται στις ίδιες προτεραιότητες και ο Αλεσάνδρο μάλιστα μίλησε προηγουμένως ε, για την σημασία της ε, εντολής που πρέπει να έχουμε. Ε, για την Κροατία ας πούμε έχουμε 113 δις εκ των οποίων ένα σημαντικό τμήμα αφορά τις επενδύσεις 24 δις ευρώ. Αυτό όμως είναι πολύ ε, λιγότερο από αυτό που δίνει κάθε τόσο σαν πίστοση ε, η τράπεζα αλλά μπορεί κανείς ε, ασφαλώς μάλλον να εκτιμήσει ότι το 25% του ΑΕΠ που, είναι, που αφορά επενδύσεις θα προωθηθεί προς τις υποδομές. Γι' αυτό λοιπόν φτάνουμε στα 8-9 δις τον χρόνο όπου το 1 δις θα είναι επιδοτήσεις και και τα 7-8 ε, θα είναι δάνεια. Ε, έρχομαι λοιπόν στο τελευταίο μου σημείο που είναι η ανάγκη ε, μακροοικονομικής, μακρόθωρης πολιτικής σε πολλαπλό επίπεδο. Ο μηχανισμός blending μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την κοινή φιλοσοφία Επίσης γνωρίζουμε ότι ήδη ε, οι τοπικές εθνικές ε, προτεραιότητες είναι συγκεκριμένες και επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική αυτή για να καλύψουμε τις ήδη δεδηλωμένες ανάγκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κανονισμό ΙΠΑ 2 αναφέρει επίσης ε, ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε, ένα, σε ισορροπία χρηματοδοτήσεων ε, σε, όσον αφορά τα project σε περιφερειακό επίπεδο όπου θα πρέπει να ε, αναλύονται οι περιφερειακές ανάγκες, οι εθνικές ανάγκες, τα συγκεκριμένα προγράμματα, η μακροοικονομική αντιμετώπιση και η μακροπρόθεσμη ε, μελέτη. Θα πρέπει όλες αυτές, ε, ε, όλα αυτά τα στοιχεία να αναλύονται από τις δικαιούχες χώρες σε συνεργασία όμως και από κοινού με τους δωρητές. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό, το έχουμε δει. Mm. Και αυτό είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ε βεβαίως ε, και ευχαριστώ που δεν εγκατέλειψα την αίθουσα και έτσι δεν είναι μια άδεια αίθουσα αυτή που όφησαν αυτή που βλέπετε στην εικόνα. Προεδρεύουσα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η μελέτη περίπτωσης για την πρώτη, για τα Δυτικά Βαλκάνια και θα δώσω τον λόγο αμέσως στον ε, κύριο ε, Κορτέσε, ο οποίος θα παρουσιάσει τον επόμενο εμπειρογνώμονα και την επόμενη παρουσίαση. Πολύ ωραία. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της Λατινικής Αμερικής. Πριν σας συστήσω τον κύριο Γκουστάβο Ερνάντες, που είναι ε, ο συντονιστής της ε, Αλόπ, να σας πω τι πιστεύει η Επιτροπή Ανάπτυξη για τη Λατινική Αμερική. Αλλά είναι η πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών της Λατινικής Αμερικής. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες σκέψεις για να καταλάβουμε την κατάσταση στη Λατινική Αμερική ε, που όλοι πολύ καλά γνωρίζετε. Από τις 18 χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι 11 έχουν αναπτυχθεί Πράγμα που τις βγάζει από τη διμερή βοήθεια. Και σε αυτές τις χώρες συγκεντρώνεται το 70% των φτωχότερων του κόσμου, παρόλο που οι ίδιες οι χώρες δεν είναι τόσο φτωχές. 73 εκατομμύρια πολιτών ζουν σε απόλυτη ένδυα στην ε, Λατινική Αμερική και 10 από τις χώρες ε, της περιοχής παραμένουν να είναι μέσα στις 15 παγκοσμίω που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανισότητες. Γι' αυτό εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή. Δεύτερον, με την ανάπτυξη και για την ανάπτυξη των χωρών αυτών και της περιφέρειας είναι πολύ σημαντικό ε, να τους βοηθήσουμε, αλλά παραμένουν πολύ ευάλωτες σε στιγμές κρίσης. Δεν είναι η ώρα να τους εγκαταλείψουμε, αλλά να δώσουμε προστιθέμενη αξία στη βοήθειά μας, που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας και τις ιδιαιτερότητες και ιδιαίτερα τις χώρες μέσου εισοδήματος, έτσι ώστε να εκριζωθεί πραγματικά η φτώχεια και να μειωθεί η ανισότητα για να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη. Εμείς τι έχουμε κάνει, τίποτα άλλο παρά να προχωρούμε στη σχέση μας με τη Λατινική Αμερική. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τη βοήθεια μας προς τη Λατινική Αμερική. Κανείς δεν θα το καταλάβαινε αυτό. Έχουμε αναλάβει πολλές δεσμεύσεις και πολιτικές και εμπορικές. Δεν μπορούμε τώρα να τους εγκαταλείψουμε. Η σημερινή χρηματοδότηση είναι 2,7 ε, δις και στην έκθεσή μου και στη διαπραγματεύσεις με τον DCI που κάνουμε, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει η συνέχιση αυτής της βοήθειας, αυτό το ποσό, με διαφάνεια και λογοδοσία. Να μπορέσουν διάφοροι τομείς να συμμετέχουν, όπως είναι πανεπιστήμια, ΜΚΟ, επαγγελματικές οργανώσεις, συνδικάτα, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ε, επιχειρήσεις και κερδοσκοπικού χαρακτήρα για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα στη Λατινική Αμερική και μέσω των ιδιαιτεροτήτων της. Η Λατινική Αμερική κατά την άποψή μου είναι το πιο εύγλωτο παράδειγμα ότι η βοήθεια και λειτουργεί και σωστά έχει γίνει και βοηθάει στην ανάπτυξη. Σώζει ζωές και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αλλάζουν οι ζωές των ανθρώπων. Και τελειώνω και θα δώσω το λόγο στη συνέχεια στο Γουστάβο Ερνάντες, τον οποίο ευχαριστώ που ήρθε. Ε, το DCI, το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας, είναι σε εμπλοκή. Είναι αδίέξοδο ο τριμερής διάλογος, χωρίς να έχει πολιτικό περιεχόμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μέσο. Και σιγά σιγά ε, ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις για άλλα μέσα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και να κατανοήσουμε επιτέλους ότι θα πρέπει να μπούμε ήδη στον πολιτικό διάλογο και να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα. Και ότι η Λατινική Αμερική θα πρέπει να είναι προτεραιότητα ως περιφέρεια για το κοινοβούλιο μας αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Και επιπλέον, αυτό δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο, όπως γνωρίζετε, κατά πλειοψηφία αποφάσισε να εγκρίνει την έκθεση για τη νέα αναπτυξιακή συνεργασία με τη Λατινική Αμερική. Αξίζει λοιπόν να σεβαστούμε στις διαπραγματεύσεις αυτά τα θέματα και να λάβουμε υπόψη την κατάσταση ορισμένων κρατών στη Λατινική Αμερική. Ιδιαίτερα αυτές τις τρεις χώρες που είναι η Κολομβία, ο Ισημερινός, το Περού ε, και από εδώ, από το Κοινοβούλιο, είπαμε ότι πρέπει να χρειαστεί διμερής βοήθεια στο μέσο αναπτυξιακής βοήθειας στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και στην έκθεσή μας υποστηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διακοπεί απότομα και να βγουν απότομα κάποιες χώρες χρειάζεται συντεταγμένη έξοδος, ένα ναι. phasing out, μια προοδευτική αποχώρηση από το πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους έτσι στη μοίρα τους. Πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό. Ε, αυτή ήταν πάει για θέση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε και ελπίζω να μπει και ένα πολιτικό περιεχόμενο σε αυτό το μέσο. Μας ανησυχεί πολύ αυτή η ολιγορία στις διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, τελειώνω εδώ εγώ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκουστάβο Ερνάντες, τον οποίο καλέσαμε, να μας κάνει ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα και εγώ να κάνω ένα σχόλιο για τα προηγούμενα, γιατί ήταν μια διαδοχή τοποθετήσεων. Δεν κάναμε ερωτήσεις. Για το blending, εγώ δεν είμαι αντίθετος. Το αντίθετο πιστεύω ότι πρέπει να το μελετήσουμε σε βάθος. Είναι ε, μια φόρμουλα που μπορεί να ε, έχει θετική έκβαση. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, χρειάζεται ένα πλαίσιο που να το ρυθμίζει αυτό με τρόπο πολύ πιο ξεκάθαρο. Αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Γιατί η συνεργασία και η ανάπτυξη δεν είναι κάτι το ξεκάρφωτο, είναι πολύ ιδιαίτερος κλάδος. Ε, θα πρέπει να ρυθμίσουμε, να έχουμε ένα πλαίσιο ρύθμισης για το blending και πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και να βρούμε ε, τρόπους και φόρμουλες να συνεργαστούμε πολύ περισσότερο γιατί εμένα με ενισχύει πάρα πολύ το εξής. Ε, όταν συζητούμε για συνεργασία ακούμε λέξεις όπως είναι αποδοτικότητα, θα βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση. Λες και αυτό μας ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, μην κάνουμε λάθος εδώ, μην συγχαίουμε διάφορα πράγματα. Άλλο είναι η προσπάθεια που κάνουμε εμείς, ε, ο δημόσιος τομέας και η κρατική χρηματοδότηση για να βελτιώνεται ε, η αναπτυξιακή βοήθεια, η διαχείριση των προγραμμάτων κτλ. Και άλλο πράγμα είναι η μαζική εισαγωγή της χρηματοδότησης και της ιδιωτικής σε προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας. Λοιπόν, και οι ιδιώτες και το δημόσιο θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι σημαντικό να βρούμε ένα κανονιστικό πλαίσιο, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο όπου να μπορούμε όλοι να το δεχτούμε και να είναι και διαφανές και αξιόπιστο. Σταματώ εδώ. Το θέτω επιτάπητος. Αλλά εγώ δεν θέλω να ιδιωτικοποιήσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Γκοστάβο Ερνάντες. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω εδώ. Είναι ο συντονιστής της ΑΛΟΠ πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών της Λατινικής Αμερικής, είναι ανθρωπολόγος, έχει πλούσιο βιογραφικό, δεν θα το αναφέρω όλο, από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Περού ε, και στα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στο ε, Μπιλμπάου και στη Βενετία διέπρεψε στις σπουδές του και στη συνέχεια πήγε στο Τέξας, στο Όστιν. Δεν θέλω να συνεχίσω το βιογραφικό σου, είναι ευρύτατο. Θέλω να σου δώσω το λόγο για να μας κάνεις την παρουσίασή σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συζήτηση αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική. Για τον εξής απλό λόγο. είναι το θέμα του blending των μεικτών μηχανισμών στην Λατινική Αμερική. Περί τίνος πρόκειται. Αυτοί οι μεικτοί μηχανισμοί μπορούν να είναι ένας ε, προνομιακός τρόπος αναπτυξιακής συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική. Εξού και η σημασία της δημόσιας συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους μικτούς μηχανισμούς και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν ως ένα νέο μέσο συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική. Έχω την πρόθεση λοιπόν στα 9 λεπτά, γιατί έχασα ένα λεπτό στην εισαγωγή μου, είναι να σας δώσω ένα συμπληρωματικό πρίσμα από την κοινωνία των πολιτών και μάλιστα από τη σκοπιά ε, μιας έρευνας που έγινε συμμετοχικής, όπως κάνουμε πάντα που συνεργαζόμαστε με διάφορους τομείς. Ένα χρόνο χρειάστηκε από τον Αύγουστο ε, του 12 μέχρι τώρα τον Ιούνιο του 13 και συμμετείχαν ε, επίσης διάφοροι ε, επιτόπου, ιδιαίτερα με αυτό το νέο τρόπο το LIFE, το Latin America Investment Facility και άλλα μέσα. Και μεταξύ άλλων είχαμε και ειδικέ συνεντεύξεις ή μη διαρθρωμένες συνεδριάσεις, εργασίας, συσκέψεις κλπ. Εδώ βλέπουμε διάφορα στοιχεία ε, και διάφορες ακροάσεις και εκδηλώσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είναι και η παρούσα ακρόαση. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι στη συμμετοχική αυτή έρευνα μπορεί να βοηθήσει στη συζήτηση και σε να συνεισφέρει η πληθώρα και η ποικιλία των ε, ενδιαφερομένων, κοινωνία των πολιτών και ε, υπάλληλοι και του Κοινοβουλίου και προσεχώς θα υπάρξει μια δημοσίευση που θα συγκεντρώσει όλες τις συστάσεις, αλλά είχαμε και εκπροσώπους και υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι τώρα αρχίζει η συζήτηση. Υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις, βεβαίως διαφορετικές απόψεις, αλλά το θέμα είναι να είναι αλληλοσυμπληρούμενες και κάπου να βοηθήσουν και να καταλήξουμε στο κοινό στόχο που είναι η βελτίωση του πλαισίου συνεργασίας. Μάλιστα. Ποια ήταν τα βασικά τώρα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Πρώτον, έχουμε αλλαγή στο ίδιο το υπόδειγμα, δηλαδή στο πρότυπο. Έχει σημασία να το τονίσουμε αυτό, γιατί είναι εφετηρία που εξηγεί όλες τις αλλαγές που έχουμε και όλο το νέο σύστημα αναπτυξιακής συνεργασίας. Δεν θέλω να επιμείνω σε αυτές τις αλλαγές, που είναι πραγματικά βαθιές αλλαγές προτύπου, παραδείγματος στο συνολικό πολιτικό τοπίο και ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να μείνω εδώ σε λεπτομέρειες, απλώς να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι βαθιές αλλαγές στη λογική την ίδια, στον ίδιο τρόπο συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ποιες είναι αυτές οι νέες λογικές αναπτυξιακής βοήθειας. Βασικά εκφράζονται από τη δημιουργία μηχανισμών καινοτόμων όπως είναι οι περίφημοι μηχανισμοί του blending. Το σημαντικό ποιο είναι να καταλάβουμε ότι η πραγματικότητα της περασμένης δεκαετίας, ετίας έχει αλλάξει εκ βάθρων. Υπάρχει μια ριζική αλλαγή που οφείλεται όπως όλοι γνωρίζουμε στην ταχεία ανάπτυξη των οικονομιών στην Λατινική Αμερική παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει η πρώτη πηγή άμεση χρηματοδότηση στη Λατινική Αμερική. Παρ' όλα αυτά το σχετικό ειδικό βάρος ε, στο εμπόριο ε, ε, πέφτει γιατί ανεβαίνουν η Κίνα κυρίως και άλλε ασιατικέ χώρε. Λοιπόν, η βασική απάντηση σε αυτό το νέο πλαίσιο ανάπτυξη που έχει αλλάξει και ριζικά καινούριο επαναλαμβάνω, είναι η ε, ατζέντα για την αλλαγή και μια νέα εστίαση στον ιδιωτικό τομέα. Τρία είναι τα στοιχεία που θεωρούμε σημαντικά στο νέο πανόραμα ε, του πλαισίου και της αναπτυξιακής βοήθειας. Μεγάλη αύξηση της εξωτερικής δράσης ως προς τους αριθμούς, Δηλαδή μεγαλύτερη εστίαση και μεγαλύτερη στήριξη του ιδιωτικού τομέα, μεγαλύτερη ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων με εγγυήσει δάνεια, κοινή ανάληψη κινδύνου και νέες μικτές ε, ε, διευκολύνσεις με το blending που είναι δωρεάν συν δάνειο. Η ατζέντα για την αλλαγή λοιπόν είναι πολύ σαφής και βασίζεται σε τρεις στόχους κυρίως υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστήριξη περιφερειακής ολοκλήρωσης και κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα για μεγάλα έργα υποδομών. Ε, νέος μηχανικός ε, LIFE, διευκόλυνση επενδύσεων για τη Λατινική Αμερική. Βασίζεται στην περιφερειακή στρατηγική για τη Λατινική Αμερική, δηλαδή ενίσχυση των στόχων στόχους ανάπτυξης για τις νέες προβληματικές των αναδυόμενων χωρών. Βλέπουμε μεγάλη αλλαγή τις τελευταίες δεκαετίες, νέα προβλήματα ε, ε, που αναδύονται, το περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και επίσης όπως υπόθηκε προηγουμένως, αυτά τα νέα στοιχεία επιζητούν να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και στα πλαίσια των δωρητών και στο διεθνές ε, σύστημα αναπτυξιακής βοήθειας. Τονίζω το βασικό στόχο της ε, Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Πολιτικής που είναι η εκρίζωση της φτώχειας. Σε αυτό το μεγάλο πλαίσιο μπαίνουν μετά από εκεί και πέρα οι επιμέρους ειδικοί στόχοι της LIFE που είπαμε ότι είναι η επενδυτική πρωτοβουλία για τη Λατινική Αμερική. Μέχρι στιγμής είναι 10 τα ε, έργα που έχουν εγκριθεί. Για να έχετε μια ιδέα, και να αρχίσουμε να προσγειωνόμαστε στην απτή πραγματικότητα. Έχουμε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα ενεργητικής απόδοσης για την Κεντρική Αμερική, ε, μικρο, με πράσινες, ε, ανανεώσιμη ενέργεια στην Ικαράγουα, ε, κλιματική αλλαγή στο Μεξικό, υδροελεκτικό εργοστάσιο στο Σαλβατόρ, Νοεμβρίου ονομάζεται. Βλέπετε εδώ πέρα όλα αυτά τα έργα να απαριθμούνται. Ένα περιφερειακό πρόγραμμα για ε, τις μεταφορές, ε, για τους εθνικούς ε, δρόμους, εθνικές οδούς στην Ήπεθρο. Το αεολικό πάρκο Κομπίνε Στύπα που είναι στο Μεξικό, είναι ένα αυτόχθονο όνομα εδώ, ηθαγενές, και επίσης στην Κολομβία η ολοκληρωμένη διαχείριση των ε, υδάτινων πόρων. Ε, βλέπετε λοιπόν όλα αυτά τα έργα και ε, τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών οργανισμών. Γνωρίζετε ποιοι είναι μεταξύ αυτών Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μαζί με κάποιους άλλους οργανισμούς από τη Λατινική Αμερική, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης και κάποιες άλλες ε, τράπεζες ολοκλήρωσης. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή λίγο στους δικαιούχους. Στο σύστημα LIFE Πώ το είδαμε από την κοινωνία των πολιτών στην έρευνα που κάναμε. Αποδέκτες είναι και οι κυβερνήσει, αλλά και τα τοπικά ή περιφερειακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εν στη Λατινική Αμερική. Και τι μας τραβάει την προσοχή. Πολλά από τα έργα που προηγουμένω ανέφερα και έχουν εγκριθεί σήμερα στη λογική του live είναι ε, έργα που εντάσσονται και σε μια προηγούμενη λογική που πολλές φορές ε, Ε, έχουν αναπτυχθεί από τις τοπικές τράπεζες και μετά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και του ελευθέρου εμπορίου. Βασίζονται σε αυτή τη λογική και πολλά από αυτά τώρα μπαίνουν στην ε, λογική των επενδύσεων από το LIFE. Θα ήθελα μόνο να σας αναφέρω δύο παραδείγματα για να αναρωτηθούμε τι είδους ανάπτυξη προωθούμε. Προηγουμένως είπαμε ότι η ανάπτυξη είναι ένα από τα βασικά και θεμελιώδη στοιχεία, για να μην πω προτεραιότητα. Όταν μιλούμε για συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική. Πολλά από τα προγράμματα αυτά στο παρελθόν προκάλεσαν σοβαρές οικολογικές ζημίες και ε, κίνησαν μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις. Να σας πω ποια είναι τα προβλήματα, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τις αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο τα θετικά, γιατί είναι τεράστια έργα. Στο 2010, ας πούμε, όπως βλέπετε εδώ, ε, στη λογική της Ήρσα, που είναι η πρωτοβουλία περιφερειακής ολοκλήρωσης της Νότιας Αμερικής ε, και χρηματοδοτείται και από το νέο πλαίσιο του LIFE. Λοιπόν, ένα τμήμα αυτών των προγραμμάτων είναι ε, διάφορα φράγματα υδροηλεκτρικά που το 2010 δημιουργήσαν μεγάλα προβλήματα στο Περού. Θυμάστε, επικυβέρνηση στο Έλαν Γκαρσία και Πρόσφατα ε, υπήρχαν ε, στον άξονα 6, εδώ στο χάρτη, ε, κοινωνικές διαμαρτυρίες στη Βολιβία, όπου πολλές ομάδες κοινωνίας των πολιτών εξεγέρθηκαν κατά της κυβέρνησης του Ιβο Μοράλες. Προσπαθούν να υπερασπιστούν προστατευμένες ζώνες των αυτοχθόνων λαών, ε, που ε, τους έχουν ε, λατήσει τη γη, εν πάση περιπτώσει κυριεύσει για την ανάπτυξη. Αυτά είναι τα βασικά έργα που υποστηρίζονται από τη μηχανισμό LIFE, οι πράσινες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις ανανεώσιμες, όπως σας είπα, μείωση του διοξιδίου του άνθρακα στο Σταλπεδόρ, ε, το υλικό πάρκο στο Μεξικό, ανανεώσιμες ενέργειες και ε, προώθηση της αιωλικής ενέργειας και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατίνων πόρων στην Κολομβία. Γιατί πήραμε αυτά τα τέσσερα παραδείγματα. Ψάχνουμε μια ισορροπία παντού, θεματική, γεωγραφική πρώτο και μετά για την κοινωνία των πολιτών και τα δίκτυα που συμμετέχουν σε αυτή τη μελέτη. για να υπάρχει μεγαλύτερη προφόρηση επιτόπου. Άλλο κριτήριο ήταν ε, η πληροφόρηση. Σε άλλες περιπτώσεις είχαμε περισσότερη πληροφόρηση, σε άλλες πιο δύσκολη και σε άλλες καθόλου, γιατί μόλις άρχισε το πρόγραμμα. Και επίσης ζητήσαμε, αναζητήσαμε και μια ισορροπία καλών και κακών παραδειγμάτων, για να έχουμε μια συλλογική διαπαιδαγώγηση όλων των ε, φορέων από το καλό ή το κακό παράδειγμα. Τελειώνω και θα περάσω στη σύνθεση τώρα. Τι διδάγματα έχουμε από την έρευνα αυτή. Πρώτον, είναι λίγη, επιπόλαιη και ε, απαρχιωμένη η δημόσια πληροφόρηση. Ε, μας κόστησε πάρα πολύ να έχουμε σωστή πληροφόρηση, παρά την καλή θέληση των διαφόρων υπαλλήλων. Μας άνοιξαν τις πόρτες τους, αλλά η πληροφόρηση που έχουν δεν είναι ενημερωμένη και δεν έχει στη διάθεση της κοινωνίας των πολιτών. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν το κριτήριο για την πρόσβαση στην ε, πληροφόρηση. Ρωτούσαμε τις τράπεζες και μας είπαν ρωτήστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά ρωτήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας είπαν αυτά τα θέματα είναι ευαίσθητα για τις τράπεζες, οπότε δεν ξέρω». Λοιπόν, όχι μόνο δεν είναι δημόσια η πληροφόρηση ούτε διαθέσιμη, παρόλη την καλή θέληση των ενδιαφερομένων, αλλά δεν υπάρχουν και πρωτόκολλα ούτε κριτήρια για το ποιο θα έχει πρόσβαση στην ενημέρωση, ποιο δικαιούται να ενημερώνεται. Και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ούτε αρμοδιότητες ούτε ευθύνε σε τελική ανάλυση. Άρα εκεί χρειάζεται και μπαίνει η διακυβέρνηση. Αν μη τι άλλο να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην ενημέρωση για να μπορούμε καλύτερα και πιο ενημερωμένοι να συμμετέχουμε στη συζήτηση. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι στιγμής από ό,τι ξέρουμε είναι παρατηρητής αυτή την πλατφόρμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα που εμπλέκεται περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρακολουθεί τους νέους τρόπους ε, συνεργασίας. Ειδικά για χώρες μεσαίου εισοδήματος. Και δεν υπάρχει πουθενά κανένας ρόλος που να προβλέπεται για τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. πολιτών. Αυτό έχει σημασία γιατί υπήρχε διακυβέρνηση στο παρελθόν, τώρα δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο, πουθενά δεν φαίνεται. Ε, δεν έχει κανένα ρόλο η συμμετοχή ε, της κοινωνίας των πολιτών. Μα μιλούμε για ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη η κοινωνία των πολιτών έχει ρόλο, γιατί έχει και γνώση και συμμετοχή και αυτό είναι θεμελιώδες άλλωστε δικαίωμα και αρχή. Συστάσεις και τελειώνω. Προηγουμένως ακούσαμε ότι τα δέντρα φαίνονται από τους καρπούς τους. Δηλαδή εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι και τα έργα μας. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη, όχι να είναι οικονομικά αποδοτικό το πρόγραμμα. Εξάντε εκ των προτέρων θα πρέπει να γίνεται ε, μία αξιολόγηση. Αν έχουμε 15 πόλεις και αυξήθηκε κατά 12% η υδροδότηση, με συγκεκριμένους δείκτες εκ των προτέρων θα πρέπει να έχουμε μια δυνατότητα εκτίμησης. Όταν κυρώνονται οι συμφωνίες σύνδεσης, να υπάρχουν μελέτες ε, αντικτύπου εκ των προτέρων, για να μπορούμε στη συνέχεια να τα αξιολογούμε. Ε, στα προγράμματα και στα έργα θα πρέπει να έχουν ενσωματωμένους μηχανισμούς ελέγχου. Ε, δεν γίνεται σήμερα αυτό και είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνουμε τα έργα. Ε, σε ποιο βαθμό κάθε έργο αποδίδει, προσφέρει και εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς στόχους με την ευρύτερη έννοια ελεύθερη και ενημερωμένη πρώτερη ε, διαβούλευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υποχρεωτικά σε όλη την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τώρα ε, τα δελτία έγκρισης των ε, έργων που δεν είναι δημόσια δεν υπάρχει δυνατότητα για μας να έχουμε πρόσβαση. Ούτε πρωτόκολλα ούτε κριτήρια υπάρχουν. Γνωρίζουμε όμως ότι σε αυτά τα μυστικά δελτία έγκρισης των σχεδίων δεν υπάρχει πουθενά κανένα κριτήριο, καμία εστίαση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ούτε στις εκ των προτέρων μελέτες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν νέα κριτήρια διαφάνειας και Λόγω δοσίας, για να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας από τους ε, φορείς επιτόπου και τέλος θέλουμε να απευθύνουμε και μια έκκληση έτσι ώστε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, εμπλακούν περισσότερο σε αυτή τη δομή της διακυβέρνησης του live. Ξέρουμε ότι τώρα είναι παρατηρητή στο Κοινοβούλιο. Η κοινωνία των πολιτών δεν έχει κανένα ρόλο ούτε στη διακυβέρνηση ούτε στην ολόκληρη τη δομή αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ Γουστάβο. Eh, Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για τη συζήτηση και θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο σε κάποιους από τους βουλευτές που είναι εδώ ενώπιον μας. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς το λόγο. Αλλά και στο κοινό. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ερωτήσεις, εάν μου το επιτρέπετε. Στον κύριο Τεβέουντε. Αναφερθήκατε στο πακέτο του blending. Στο μέλλον η κάθε μία οργάνωση θα κάνει ε, το, ένα τμήμα ας πούμε του πακέτου ή όλοι μαζί όλο το πακέτο. Δεύτερον για τα Βαλκάνια στους δύο εκπροσώπους ε, της ε, Κεντρικής ε, Τράπεζας. Βλέπετε, θεωρείτε το blending στα Δυτικά Βαλκάνια να είναι πιο εύκολο να επιτύχει από ότι σε άλλες περιοχές. Δεύτερον, σε ποιες περιπτώσεις δεν λειτουργεί το blending. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Ριβέλε. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν είναι όμως εύκολη απάντηση. Εξαρτάται από τις περιστάσεις αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες από τη μεριά των υποδοχέων ε, έχουν όλο και περισσότερες επιλογές μεταξύ διαφόρων μορφών ε, ε, χρηματοδότησης. Είναι η λεγόμενη age of choice, είναι η εποχή των επιλογών. Και επομένως αυτό το λαμβάνουν υπόψη τους οι αναπτυσσόμενες χώρες, αν μελετούν, βλέπουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε πηγής αυτό που νομίζω πως είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμό σίγουρα. Εάν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ένας οργανισμός να ασχοληθεί μονάχα με το συντονισμό, τότε ναι, μας το κάνει. Κάθε, κάθε οργάνωση, κάθε θεσμικός φορέας όμως μπορεί να δώσει το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Αυτό που, σημαίνω είναι, αυτό που θέλω να εννοήσω είναι ότι ε, όλες οι πηγές ε, θα πρέπει να συνενωθούν. Θα, όπως βάζουμε τα δάνεια μαζί με τις επιδοτήσεις, θα πρέπει και οι φορείς ε, να εμπλέκονται σε στενή συνεργασία. Να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου ο καθένας θα αναλαμβάνει να φέρει εις αυτό που γνωρίζει καλύτερα και επομένως θα πρέπει να υπάρχουν ήδη τα εργαλεία τα οποία ο καθένας την κατάλληλη στιγμή θα μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ε, κάθε φορά δηλαδή να επιλέγει ποιον πόρο, ε, με ποιο τρόπο. Ε, να, να αποφασίσουν δηλαδή ποιος αποφασίζει για πόσους πόρους, για ποιους, για πόσο μεγάλο διάστημα κτλ μεγαλύτερο συντονισμό, όχι μονάχα μεταξύ των επιδοτήσεων και των δανείων, αλλά και των εμπλεκομένων φορέων. Καλύτερος, αποτελεσματικότερος συντονισμός. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο, ο διάδρομος βορρά-νότου. όπου διαφορετικοί φορείς έχουν ε, εμπλακεί και βλέπουν πώς από κοινού μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δεσμευτικές υποχρεώσεις. Ε, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί τεχνική βοήθεια, σε άλλες περιπτώσεις ε, χρηματοδοτική πόρη και με αυτόν τον τρόπο είναι καταλητική η συμμετοχή όλων. Βεβαίω, καμιά φορά μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου συντονισμού μπορεί να υπάρχουν κάποιες κόχες, κάποιες νήσες καλύτερης, μεγαλύτερης συνεργασίας ανάμεσα σε δύο ε, οργανώσεις ή δύο ε, φορεί. Ελπίζω να απήντησα στην ερώτησή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεβέλε. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Καράνο τώρα. Σας κατευχαριστώ για το ερώτημα για τα ερωτήματα. Θα απαντήσω στο πρώτο, κατά πόσον δηλαδή ο σχεδιασμός είναι στην Ευρώπη είναι πιο επιτυχής από ό,τι αλλού. Δεν είναι εύκολο να εύκολη απάντηση, εξαρτάται από τα κριτήρια της επιτυχίας. Έχουμε δει τα δεδομένα για τη μόχλευση και τα ποσά των δωρεών που έχουν χορηγηθεί σε σύγκριση με τα δάνεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τεράστια διαφορά για αυτούς τους δείκτες. Υπάρχουν όμως και μερικές διαφαρές που σχετίζονται με τα διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια της Ένωσης. Εμείς λειτουργούμε υπό την ενωσιακή πολιτική, άρα αναπεριφέρεια. Στα Δυτικά Βαλκάνια συγκεκριμένα τονίζουμε, τονίζεται ιδιαίτερα η σύγκληση προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τονίζεται ιδιαίτερα η ιδιοκτησία από τους ωφελουμένους μετά ιδίω την μελλοντική τους ένταξη. Αυτό οδηγεί σε ορισμένες διαφορές. Δεν θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένο το πρότυπο αυτό, αλλά είναι ένα βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τον σχεδιασμό. Και η ιδιοκτησία βέβαια είναι σημαντικό κριτήριο και γι' αυτό μουτά της μουτάντης είναι αρχή που το, συζητάμε αυτή τη στιγμή στην οργάνωσή μας. Άλλο στοιχείο διαφοροποίησης είναι η δυνατότητα στα Δυτικά Βαλκάνια που είναι λιγάκι περισσότεροι να χρησιμοποιούνται δωρεές και από άλλους, από μη Ευρωπαίους δωρητές όπως το Καναδά, την Νορβηγία. Και όλα αυτά διαφοροποιούν την κατάσταση. Είναι σημαντικό νομίζω να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε αυτά και σε άλλες συνθήκες όποτε μπορούν να συμμετάσχουν μη Ευρωπαίοι δωρητές. που είναι και η πιο δύσκολη και σπάνια πηγή χρηματοδότησης που έχουμε. Υπάρχει για το θέμα της πολιτικής θέλησης το έθεσε πρώτη φορά το Συμβούλιο που απέτησε απλοποίηση των διαφόρων εργαλείων που αρχικά είχαν προτείνει οι ίδιοι ωφελούμενοι. Στη Μεσόγειο γενικότερα υπάρχει από τη μια μεριά ένας ενιαίος μηχανισμός blending αλλά υπάρχουν και λειτουργούν και άλλα μέσα όπως τα ταμεία Ντοβίλ κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ή να απορροφηθούν περισσότερα σε ένα ενιαίο πλαίσιο για συγκεκριμένες περιφέρειες όπως τη Μεσόγειο. Για το δεύτερο ερώτημα τώρα. Δύσκολο και αυτό, πολύ δύσκολο. Αλλά να κάνω μερικά σχόλια. Καταρχήν, το blending σε κάποιο βαθμό είναι και θέμα κοινή λογικής τουλάχιστον αν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος ο ενωσιακός προϋπολογισμός να κινείται προς διαφορετική κατεύθυνση από ότι τα ενωσιακά δάνεια. Είναι λογικό λοιπόν να συνδυαστούν οι πόροι που διαθέτουμε είτε είναι δωρεές είτε είναι δάνεια και δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι το καλύτερο. Σίγουρα είναι λιγότερε οι δωρεέ για διάφορου λόγους και τα δάνεια επίσης είναι περιορισμένα αλλά ίσως να μπορεί κανείς να είναι πιο ευέλικτο με τα δάνεια. Είναι θέμα βαθμού. Λογικό είναι λοιπόν να συνδυαστούν με τις σωστές προτεραιότητες. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία της επιλογής προτεραιοτήτων θα ήθελα να τονίσω ότι στα Δυτικά Βαλκάνια χρηματοδοτούμε κυρίως τον δημόσιο τομέα, προγράμματα του δημόσιου τομέα, αν και αφήνουμε λίγα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Αλλά τα κυριότητα περισσότερα είναι για το δημόσιο τομέα. Εδώ λοιπόν που επιλέγουμε τα χρήματα που θέλουμε να διαθέσουμε υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν λειτουργούν τα πράγματα γιατί εξαρτάται από το μέλλον ενός σχεδίου η αποδοτικότητά του. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι να έχει κάνει κανείς λάθος από την αρχή, αλλά ίσως είχε αξιολογηθεί λάθος η επένδυση, ίσως ε, το ποσό δεν αρκούσε, μπορεί, μπορεί πολύ να είναι οι λόγοι. Αλλά προσπαθώ να σας απαντήσω σε σύγκριση με την παρουσίασή μας ότι δηλαδή δεν λειτουργεί το πράγμα όταν υπάρχει μία δωρεά τεχνικής βοήθειας και βάζετε χρήματα στην προετοιμασία του σχεδίου αλλά το σχέδιο δεν εφαρμόζεται ποτέ. Εκεί σαφώς τα χρήματα δεν έχουν σωστά δαπανηθεί γιατί δεν πετύχατε το αποτέλεσμα που θέλατε την αύξηση δηλαδή της παραγωγικής τα κτλ. Σε πιο μικροσκοπικό επίπεδο μπορεί να υπάρχει περίπτωση να θεωρήσει κανείς ότι πάλι δεν λειτουργεί το πράγμα αλλά μπορεί να είναι και η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος ας πούμε μερικοί από τους ισχύοντες κανονισμούς μπορεί να είναι να αναγκάζουν την εφαρμογή ορισμένων προγραμμάτων. Βέβαια δεν είναι στόχος μας να επηρεάσουμε τους πολιτικούς, αλλά θέλουμε να συνδυάσουμε το μακροεπίπεδο με το μικροεπίπεδο. Το τελευταίο αυτό σχετίζεται με το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και σε, κάποια, σε κάποιο βαθμό πρέπει να αφήσουμε κάποιο περιθώριο για την επιτυχία των προγραμμάτων. Αυτό ήθελα να σας πω, να αυτό. αυτό. Σας ευχαριστούμε κύριε Συγκολάνη. Η κυρία Νίμσκι μήπως θέλει να μας βγάλει κανένα συμπέρασμα. Mm. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Κορτές, ευχαριστώ συνάδελφοι. Νομίζω ότι πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν το απόγευμα και θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ε, το πλέον προσήκον μέρος έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Έχω σημειώσει κάποια στοιχεία. Το blending δεν είναι μηχανή που βγάζει λεφτά αλλά μπορεί να εκπομπή πάρα πολύ χρήσιμο. Δεύτερο σημείο, τα, οι μηχανισμοί μόχλευσης ε, είναι σημαντικά, σημαντικοί, αλλά δεν είναι πολύ σαφές ακόμα ποιος μοχλεύει τι και αν όλα αυτά, ε, όλες αυτές οι προσπάθειες ε, είναι καλά προσαρμοσμένες στην ε, παρούσα κατάσταση και στις ε, ανάγκες ε, των δικαιούχων. Να μην λησμονούμε επίσης ότι ο συντονισμός των δωρητών είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της αύξησης της αποτελεσματικότητας και επομένως ο συντονισμός μεταξύ τους πρέπει να αυξηθεί είτε υπάρχει το blending είτε όχι. σε σχέση με τα καινοτόμα ε, εργαλεία. Πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν έτσι ώστε να καταλάβουμε ακριβώς με ποιο τρόπο όλα, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί μπορεί να μας οδηγήσουν σε καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση μέσα από συνεδριάσεις σαν αυτή που είχαμε σήμερα. Θα συνεχίσουμε βέβαια και την ανταλλαγή ε, των απόψεων και θα συνεχίσουμε με τη δημιουργία σωστών ε, ε, πρωτοβουλειών. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και είμαι βεβαία ότι και στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιλήσουμε σοφία από την πραγματογνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ.